So, good, good morning, colleagues. Καλημέρα συνάδελφοι. Καλώ ήρθατε στη συνεδρίαση. Πρώτο σημείο. Έχουμε δύο θέματα. Τι Ευρωπαϊκού παρόχους υπηρεσιών πληθοπορισμού, επιχειρήσεις και επίσης και τις αγορές ε, για τα χρηματοστικά μέσα. Λοιπόν, από τέσσερα λεπτά έχουν οι σκιώδεις, έξι οι ε, εισηγητές και θα δώσουν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον πληθοπορισμό, το ECSP για την υπηρεσία, δηλαδή παροχή πληθοπορισμού για τις επιχειρήσεις, ε, έχει το λόγο Ashley Fox. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους. Έτσι, μπορέσαμε να τηρήσουμε το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα με καθησυχάζουν και οι τροπολογίε και οι διεξαχθεί ε, συζητήσει με τους κοιόδης. Πιστεύω ότι κινούμεθα προ την ίδια κατεύθυνση και πολλά από τα θέματα μέχρι τώρα δεν ήταν επίμαχα. το χάρη, αύξηση στα 8 εκατομμύρια του ορίου του πληθοπορισμού και ε, αύξηση της προστασίας των επενδυτών. Όλοι, όλες οι ομάδες υποστηρίζουν αυτές τις προσεγγίσεις. Τρεις τομεί εντοπίσαμε όμως, όπου δεν υπάρχει ομοφωνία και θέσα τα σχόλιά μου να, αφορούν, να αφορούν τους τρεις τομείς. Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΣΜΑ, η συμπερίληψη των ε, ICOs και το καθεστώς τριών ε, ε, τρίτων χωρών. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το ρόλο της ΕΣΜΑ και προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ΕΣΜΑ να αδειοδοτεί και να υποπτεύει τις πλατφόρμες πληθοπορισμού αλλά αρκετοί σκιώδεις είναι πιο διστακτικοί για το θέμα αυτό εμού συμπεριλαμβανομένου. Η άποψή μου είναι ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές είναι σε καλύτερη θέση να κατανοήσουν ποιες είναι οι αποχρώσεις που επικρατούν στις αγορές τους και να έχουν ορθή διακυβέρνηση των πλατφορμών που λειτουργούν εκεί. Αυτός ο κανονισμός ε, εξαρτάται από την εξασφάλιση ότι χρησιμοποιείται η αδειοδότηση ενδεδειγμένη και επίση ακολουθούνται οι αρμόδιοι κανόνε για το καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο. Η υποπτή γίνεται σε εθνικό επίπεδο και έτσι θα μπορούσε η υποπτική επίβλεψη τη ΕΣΜΑ να περιοριστεί, αν ζητήσουν την ΕΣΜΑ να ασκήσει αυτή ε, τον έλεγχο σε αυτό το τομέα. Και δεν έχει αρκετού πόρου η ΕΣΜΑ να μπορεί να διοδοτεί και να υποπτεύει το καθεστώ αυτό. Χθε είχαμε τους προέδρους των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών που ήρθαν να μιλήσουν στην Επιτροπή και έθεσα το θέμα της αρμοδιότητας προς τον Στέβεν Μαϊόρ που ήταν ο πρόεδρος της ε, ΕΣΜΑ. Ε, καλωσόρισα την απάντηση που έδωσε. Είπε ότι δεν θα είχε νόημα να δώσουμε δραστηριότητες μικρότερης κλίμακας στο φορέα που δεν ανήκουν αποκλειστικά στην Ευρώπη, στις εθνικές αρμόδιες αρχές και εμπλέκουν μόνο την ΕΣΜΑ όταν αυξάνεται η κλίμακα. Ε, 8 εκατομμύρια ευρώ είναι το ανώτατο όριο αυτού του καθεστώτος. που δεν θα μπορούσε αυτό να θεωρηθεί ότι είναι συστημικά σημαντικό ποσό. Τι προσπαθούσε να πει ο πρόεδρος της ΕΣΜΑ. Ότι αυτό θα έπρεπε να το αφήσουμε στις εθνικές αρμόδιες αρχές. Και προσβλέπω στις ε, συζητήσεις που θα ακολουθήσουν το απόγευμα επ' αυτού. Δεύτερο θέμα, η συμπερίληψη των ICOs. Αυτό δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα δυναμική όπου οι απόψεις των σκιωδών και των ομάδων τους ε, δεν ε, θυγραμμίζονται πάντα. Οι τροπολογίες μου που υπευλήθησαν μαζί με άλλους συναδέλφους από διάφορες ομάδες όπως από το ΕΛΚ και από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες προσπαθούν να αποσαφηνίσουν κάτι ότι αν είναι μια πλατφόρμα Ισχύει αυτό που λέω όταν μια πλατφόρμα συμμορφώνεται τα εξή. Δηλαδή σε πλατφόρμες όπου πρώτα απ' όλα Μήπως θα μπορούσαν να σταματήσουν κάποιες συζητήσεις, να έχω ησυχία. Ησυχία, λέει ο Πρόεδρος, παρακαλώ, ησυχία. Λοιπόν, πρώτον, λέει και ο Άσλε Φόξ, όπου έχουμε κεντρικό εκδότη που μπορεί να λογοδοτεί για το πρόγραμμα που προσφέρετε. Δεύτερον, χρησιμοποιείται ενδιάμεσος για να εκδώσει τα αρμόδια έγγραφα και δεν είναι ιδιωτική τοποθέτηση. Τρίτον, εκδίδει έγγραφα προσφέροντας ένα δάνειο ή ε, διάφορα αξιόγραφα που μπορούν να μεταφερθούν και τέταρτον η διαφορα αξιογραφα που μπορουν να συνάδει με τις ε, διατάξεις του κανονισμού. Δηλαδή η προσφορά είναι κάτω από τα 8 εκατομμύρια ευρώ και τότε και μόνο τότε θα συμμορφούνται με τον τρέχοντα αυτό, με τον ισχύοντα κανονισμό. Τούτων λεχθέντων, πολλοί σκιώδεις είπαν ότι δεν θεωρούν ότι αυτή είναι η σωστή έκθεση που θα ε, διευθετεί αυτές τις πλατφόρμες. Ε, Κατανοώ τις ανησυχίες και συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι ένας κανονισμός στα μέτρα του τομέα θα πρέπει ε, να υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι ό,τι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορέσει να ετοιμάσει μια πρόταση όμω, θα είναι πολύ αργά δοθήσει τη ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η αγορά. Ε, Αυτό ο κανονισμό αποτελεί τέλεια ευκαιρία να τονίσουμε το πώ κάποιε πλατφόρμες μπορούν να συμμορφωθούν με αυτόν τον κανονισμό και να καθορίσουν εθελοντικά πρότυπα με τα οποία θα μπορούν να συμμορφωθούν για να αποκτήσουν ε, νομιμοποίηση και θα μπορούν να γίνει, θα μπορεί να γίνει ένα διαχωρισμός των προγραμμάτων τα οποία είναι νόμιμα από τα παράνομα. Τελευταίο θέμα, Πρόεδρε, είναι το καθεστώς για τις ε, τρίτες χώρες ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι επανυποβάλλατε εκείνα τα τμήματα των τροπολογιών μου, της εκθέσεώς μου, υπομορφή τροπολογιών. Πιστεύω ότι το άρθρο που προτείνω επιτρέπει την εξαγωγή των βελτίστων πρακτικών και ενθαρρύνει τη διεύρυνση της αγοράς που δεν γνωρίζει σύνορα πέρα από την ενιαία αγορά και οδηγεί στι νεοφυεί επιχειρήσει, μικρομεσαίε επιχειρήσει να αποκτήσουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ε, προβληματίστηκα από την αντίδραση που προβλήθηκε σε αυτή την ιδέα. Εγώ ζητώ αυτό το καθεστώ να επιτρέπει σε τρίτε χώρε που υθετούν αυτό τον κανονισμό εξ ολοκληρού για τι πλατφόρμες που θέλουν να έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά ε, να μπορούν να αναγνωριστούν σαν ισοδύναμες υπηρεσίε. Οι τροπολογίε μου μιμούνται το καθεστώ βαθμολόγηση και αναφέρουν ε, και κάποια σημεία τα οποία αναφέρει στην έκθε... αναφέρονται στην έκθεση Hayes. Κάποιοι σκιώδεις ακόμα δεν ενδιαφέρονται στο να συζητήσουν το θέμα. Και τι υποθέτω από αυτό. Ότι εμπλέκεται η πολιτική ε, πολιτική απόχρωση επηρεάζει αυτέ τι αποφάσει και όχι η ορθή λογική για τι σωστέ πολιτικέ αποφάσει. Χαίρομαι πολύ μέχρι, τούδε ε, την τούδε επιτευθύσα πρόοδο και προσβλέπω στι συνομιλίε με του Σκιώδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσλι. Επόμενο εισηγητή για, το, για τι αγορέ και τα χρηματοσυντικά εργαλεία. Η Κάρα Νατιγκάλη δεν είναι εδώ. Ο Ραμόν θα μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ζητά συγγνώμη η Καρολίνα που απουσιάζει και γι' αυτό μου έστειλε κάποια σημείο στο θα διαβάσω. Ευχαριστεί λοιπόν τον Άσλεϊ και όλους τους κοιόδης για την καλή συνεργασία στις συνεδριάσεις και προσβλέπει σε περαιτέρω συζητήσεις επόμενες εβδομάδες. Η Καρολίνα επίσης ευχαριστεί τους συναδέλφους για τις νέα τροπολογίες που υπευλήθησαν στην έκθεσή της. Οι τροπολογίε που υπέβαλε η Καρολίνα για την έκθεση του Άσλε έχουν σαν στόχο τη βελτίωση τη συμμετοχή των εθνικών αρμοδίων αρχών υποστηρίζει την, να συμπεριλαμβάνεται να μειωθεί το όριο και έτσι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να αφεληθούν από το νέο καθεστώς. Η αύξηση του ορίου και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή φαίνεται ότι είναι κάτι που δεν δημιουργεί προβλήματα για αυτήν. Όμως ε, πιο δύσκολη είναι η συμπερίληψη των αρχικών προσφορών νομισμάτων που προτείνεται και μια αναθεώρηση κατά χώρα και συνεργασία μεταξύ της ΕΣΜΑ και των Εθνικών Αρμοδίων Αρχών. Η Καρολίν επίσης καλωσορίζει τις φιλόδοξες απόψεις του Άσλεϊ και κάποιων συναδέλφων μας ε, και συμφωνεί μαζί τους και μια ταχεία έγκριση μιας νομοθεσίας που διευκολύνει ε, την, τα κρυπτονομίσματα και τα νέα νομίσματα είναι ύψης της σημασίας. Ε, γι' αυτό παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μια πλήρη αξιολόγηση ενδεχομένου νομικού πλαισίου για το νέο, για το νέο αυτό τρόπο χρηματοδότησης νοφιών επιχειρήσεων και αύξηση του μεγέθους επιχειρήσεων και να αποφύγουμε κάθε καθυστέρηση από αυτού. Όσον αφορά την ΕΣΜΑ και τις Εθνικές Αρμόνες Αρχές υποστηρίζει τον βελτιωμένο ρόλο των Εθνικών Αρμοδίων Αρχών διότι αυτές οι αρχές είναι αυτές που ξέρουν τις αγορές με τον καλύτερο τρόπο. Όμως διαφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αφαιχτούν διότι αυτό είναι περίπλοκο, και αυτό είναι περίπλοκο θέμα για συμβιβασμούς. Η διατάξη τη χώρε φαίνεται να γίνεται το δύσκολο θέμα τη θητεία αυτή και σε, αναδύεται σε κάθε χαρτοφυλάκιο και πάντα είναι επίμαχο το θέμα. Θέλουμε τελικά να υποστηρίξουμε διαφάνεια, ανοιχτέ αγορέ και φιλόδοξε διατάξει ε, ισοδυναμία. Παρόλο που αναγνωρίζουμε την πολιτική ευαισθησία του θέματο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκέ μικρομεσαίε επιχειρήσει να μπορούν να χρηματοδοτούνται είτε αγέντα αυτό από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο είτε από αλλού. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ραμόν. πάμε στους σκιώδεις. Δύο σκιώδεις του ΕΛΚ. Αν Σάντερ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και την, τον συγητή και τις σκιώδεις συγητές για τις ε, καλές ε, συναντήσεις που είχαμε και τη συνεργασία και που θα έχουμε και στο μέλλον. Δύο πράγματα. Πρώτον, το θέμα των ορίων συμφωνώ με τους συναδέλφους μου, την πλειονότητά τους. Θέλω να αυξηθεί το κατώτατο όριο για τη δημοσίευση ε, του προσπέκτου στο βασικό εγγράφου πληροφοριών από 1 εκατομμύριο σε 8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά την προστασία των επενδυτών, νομίζω ότι χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ενδεχόμενοι ε, επενδυτές να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα και στις προσφορές της. Αυτή τη στιγμή έχουν δώσει κάποιες πληροφορίες, όπως οι προσωπικές ε, πληροφορίες και να έχουν δώσει ε, μια εξέταση γνώσεων, να έχουν δώσει εξετάσεις, δεν να έχουν περάσει εξετάσεις, να αποδεικνύουν ότι είναι ενήμεροι και έχουν λάβει και τις προειδοποίησεις της πλατφόρμας σε περίπτωση που ε, δεν ε, γνωρίζουν αυτά τα θέματα. Τώρα, σε σχέση με τα έργα που προτείνονται. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι πλατφόρμες που θέλουν να επενδύσουν στα προτινόμενα έργα να μπορούν να το κάνουν. Είναι το περίφημο skin in the game, δηλαδή όταν έχεις κάτι ε, που διακυβεύεται στο συγκεκριμένο θέμα, ε, έχεις κάτι να χάσεις. Δεν είναι όμως συστηματική υποχρέωση αυτή, απλώς χρειάζεται καλή ε, ενημέρωση των επενδυτών. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να είναι διαφανή η πλατφόρμα και να κάνει καλή ενημέρωση. Θα πρέπει να γίνεται επίσης μια διάκριση ανάμεσα στην ε, πληροφόρηση προς το κοινό της πλατφόρμας και την επικοινωνία, το marketing, τη διαφήμιση που απευθύνεται στους ε, καταχωρημένους επενδυτές στην ίδια την πλατφόρμα. Και έρχομαι στα τρία πιο προβληματικά τώρα θέματα, euh, στα οποία χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Το πρώτο είναι το θέμα της εποπτείας. Τώρα, δημιουργούμε ένα ευρωπαϊκό μέσο και κατά την άποψή μου θα ήταν ενδιαφέρον και σκόπιμο η ε, άδεια η ε, έγκριση και η εποπτεία να ανατεθεί στην ΕΣΜΑ, την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Κατανοώ τα αντεπιχειρήματα, το θέμα των αρμοδιοτήτων κτλ. Αλλά Ας έχει αυτή την αρμοδιότητα η ΕΣΜΑ και από εκεί και πέρα και ε, οι εθνικές αρχές θα τις εκχωρήσουν τις αρμοδιότητες αυτές. Παραμένει ένα θέμα μετά τη συζήτηση που είχαμε στην ομάδα μας που έχει ενδιαφέρον να μάθουμε την ε, νομική γνώμη, τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε να αναθέσουμε αυτή την αποστολή στην ΕΣΜΑ ε, γνωρίζοντας ότι αυτό σήμερα δεν προβλέπεται στις αρμοδιότητές της. Γιατί επίκειται και η αναθεώρηση ε, των οργανισμών αυτών. Εμείς μπορούμε τώρα να τις αναθέσουμε τέτοια καθήκοντα πριν την αναθεώρηση. Επόμενο θέμα. Το σύστημα ισοδυναμίων. Γνωρίζουμε σήμερα ότι θέλουμε να αναπτύξουμε αυτή την αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είμαι βέβαια. για το ποιο είναι ο στόχος. όλων. ο δικός μας στόχος είναι να αναπτυχθεί η αγορά του crowdfunding στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τελευταίο που αφορά ε, στην αρχική προσφορά νομισμάτων, συμφωνώ με κάποιους συναδέλφους, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται οπωσδήποτε ρύθμιση και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει προτάσεις. Από την άλλη όμως, πιστεύω ότι το κείμενο για το crowdfunding δεν είναι τώρα το κατάλληλο νομοθέτημα για να ρυθμίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά. Και θα χαρώ να δω τις συζητήσεις που θα ακολουθήσω τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, uh, for contribution and... Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβαση. Ο Τόμ τώρα θα μιλήσει εκ μέρους του ΕΛΚ, σαν εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι σαφές νομίζω πλέον ότι η συζήτηση για τα εικονικά νομίσματα ε, βγήκε στην επιφάνεια και για αυτό το θέμα. Το είπε και η συνάδελφος Σάντερ, εκτός ε, από τα άλλα θέματα που μας έχουν τραβήξει την προσοχή. Ε, τώρα να τα βάλουμε όμως σε μια σειρά. Πρώτον, υπάρχουν διαφορές και είναι και μεγάλες ανάμεσα στο ρυθμισμένο crowdfunding και ε, από την άλλη τα ICO. 8 ε, εκατομμύρια ευρώ αναφέρθηκε ε, το ποσό το κατώτατο για το crowdfunding. Είναι πολύ μικρό λοιπόν το κλάσμα των ICO που θα καλυφθεί της αρχικής κυκλοφορίας κάποιων νομισμάτων. Επίσης, ε, σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει δυναμικό ε, ανάπτυξη των εικονικών νομισμάτων, αλλά δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να τα ρυθμίσουμε ακόμα. Είναι πολύ λίγη γνώση που έχουμε και η Επιτροπή μας και εγώ θα ήθελα να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη ενημέρωση και πληρέστερη έτσι ώστε να ε, δούμε ξεχωριστά το θέμα των εικονικών νομισμάτων και όχι εμπαρόδο τώρα στο crowdfunding και πάλι για τα εικονικά ε, νομίσματα. Βεβαίω δεν μπορούμε εμεί να μείνουμε στο περιθώριο. Στην Ασία είναι πάρα πολύ δημοφιλή αυτά. Δεν σημαίνει ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να αδρανίσουμε. Βεβαίω χρειάζεται ρύθμιση και προστασία των καταναλωτών. Ε, αυτό είναι δική μας δουλειά. Από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να ε, στραγγαλίσουμε και την αγορά και να την αφήσουμε να ε, πεθάνει. Αυτό είναι ένα νέο ε, λουλουδάκι, τα εικονικά νομίσματα που θα πρέπει να του νερό και οξυγόνο για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να μην μαράθει. Αυτά από τη πλευρά της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Τόμ. Από τους σοσιαλιστές, Καϊλή. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον Ασλέ και τους συναδέλφους που πάνω στο θέμα. Συγχαρητήρια για την πρόοδο. Συμφωνούμε μάλλον επί του βασικού αντικειμένου. Τα 8 εκατομμύρια δηλαδή ως α, Συμφωνήσαμε για τους ορισμούς λίγο πολύ. Συμφωνούμε με τις συμβαστικές για την διαχείριση παραπώνων, την ενημέρωση των πελατών, την αποκάλυψη των ποσοστών αφαίρεσης κλπ. Όσον αφορά τις αρχικές προσφορές νομισμάτων, εγώ θα ήθελα να τους περιλάβουμε στο θέμα, να βρούμε τώρα με ποιον τρόπο ακριβώς θα γίνει αυτό, για να έχουμε και ένα πλαίσιο νομικής ασφάλειας, για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές σε ένα άγριο περιβάλλον πριν είναι πολύ αργά μπορούμε να συμπληρώσουμε το πλαίσιο. Όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, η θέση μα είναι ότι το κείμενο της Κομισιόν ε, είναι καλό. Το πνεύμα του νομοθέτη δεν είναι να υποκραστήσει τι εθνικέ αρχές με την ΕΣΜΑ, αλλά να δημιουργήσει ένα ομογενέ περιβάλλον, ειδικά στι χώρε που δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο για τον πληθυπορισμό. Και ε, γι' αυτό το λόγο δεν Καταλαβαίνω γιατί το προτείνεται ένα διαφορετικό καθεστώς. Όταν είναι σαφές ότι η Ένωση Εταιριών Πληθυπορισμού προτιμούν αυτό που λέει και η Κομισιόν εν τέλει. Τέλος, ευχαριστώ τον Ashley Φόξ για την προσπάθεια του να βρει λύση όσον αφορά την ισοδυναμία εναντί τρίτης χώρας. Πρόκειται για κανονισμό για τα κρατημέλη, έτσι, αυτό θυμίζω. <laughs> Δεν μιλάμε για τις τρίτες χώρες εδώ, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο κείμενο. Μπορούμε να βρούμε μια λύση γι' αυτό αργότερα. Όμως σε αυτή τη φάση ε, δεν συμφωνούμε με το προτινόμενο άρθρο. Αυτά από εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Εύα. Και τώρα, από τους πράσινους, μόλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Ashley και τους βοηθούς του για το εξαιρετικό πόνιμα. Να σου πω πού συμφωνούμε. Συμφωνούμε με την πρωτοβουλία για την ενιαία πλατφόρμα. Θα δούμε την ορολογία ακριβώ, αλλά με την αρχή συμφωνούμε. Σίγουρα θα διευκολυνθεί η εναλλεκτική χρηματοδότηση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και άλλες επιχειρήσεις. Ε, όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών, βλέπω να γίνεται μια κίνηση. Νομίζω πήγαμε καλά με τις συμβαστικές τροπολογίες. Όλοι όμως οι σκιώδεις ε, επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες, για παράδειγμα ισοδυναμία με τρίτες χώρες. Η θέση μας είναι ότι δεν πρέπει ακόμη να δημιουργήσουμε ισοδυναμίες στην αγορά πληθοπορισμού, γιατί είναι μια καινούρια αγορά, μια νεοφυής αγορά, ακόμη και σε εμά, ε, παρά το γεγονό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προηγείται, είναι μπροστά σε αυτόν τον τομέα, αλλά ε, νομίζω ότι είναι πολύ ε, να προχωρήσουμε αυτές τις ισοδυναμίες. Όσον αφορά την εποπτεία και τις σχετικές αρμοδιότητες. Νομίζω ότι πρέπει, η ΕΣΜΑ πρέπει να είναι επικεφαλής εδώ και να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ ΕΣΜΑ και των εθνικών αντιστοίχων αρχών. Για τα SEO, στι αρχικέ προσφορέ νομισμάτων, είμαστε κοντά στο ΕΛΚ. Δηλαδή, αντί να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε ένα μικρό κομμάτι μόνο αυτή τη αγορά ε, από σπόντα μέσω άλλου τρόπου, καλό θα είναι η Κομισιόν να υποβάλει ένα ειδικό νομοθέτημα για να καλύψουμε και αυτό το θέμα. Εδώ λοχεύουν πολύ σημαντικοί κίνδυνοι και χρειάζονται χρειάζεται να εμπλακούν οι ειδικοί, πραγματικά ειδικοί από κάθε χώρα. Ο εισηγητή επίση είπε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ πολιτικών ομάδων για να πάμε στα 8 εκατομμύρια. Όμω, εγώ το είπα στου Κιώδη ότι δεν θα συμφωνήσουμε τα 8. Χρειάζεται μια προληπτική προσέγγιση να το κρατήσουμε στα, στο 1 εκατομμύριο. Αυτή είναι και η θέση μας. Και είναι κρίμα γιατί είδα πολλέ τροπολογίε μα δεν έχουν συμπεριληφθεί, δεν έχουν ενσωματωθεί στι συμβαστικέ, ειδικά η 249 για τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει, για τι πλατφόρμε πληθοπορισμού. Είναι παρόμοια τροπολογία με του σοσιαλιστέ. Ελπίζω ότι θα περάσει, θα έχει πλειοψηφία. Και η 282, ανταλλαγή έλεγχο που πρέπει να γίνει όσον αφορά του κυρίου των έργων. Θα ξαναπούμε βεβαίω οι σκιώδει, έχουμε σκέψει μπροστά μα πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ικανές συμβαστικέ τροπολογίε. Βάσει το στο πνεύμα από την δεν είναι κανείς εδώ, άρα η ευθύνη ε, Μαρκο Βάλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ και το συγητή και το σκιώδη συγητή για την ανταλλαγή απόψεων και βρήκαμε κάποια σημεία συμφωνίας και χαίρομαι που βρήκαμε μια συμφωνία όσον αφορά το όριο από 1 στα 8 εκατομμύρια ευρώ περιορισμοί που πρέπει να μπουν ε, για το λιανικό εμπόριο, για, το, για την πλατφόρμα αυτού του πληθοπορισμού πρέπει να ευθυγραμμιστούν ε, σωστά με τους κανόνες, κάποιο περιορισμό στην απαγόρευση επενδύσεις για τους ε, εξαρτώμενους εργαζομένους, υποχρέωση να δημοσιεύεται το rate of default των διαφόρων προγραμμάτων των πλατφορμών και καλύτερα να αποφευθούν συγκρούσεις ε, συμφερόντων και επικρατεί μεγαλύτερη διαφάνεια με αυτόν τον τρόπο. Επ' αυτών των σημείων συμφωνήσαμε και μέχρι τώρα είχαμε μεγάλη επιτυχία. Έχουμε τρία σημεία που πρέπει να απεμπλακούν για την συμπερίληψη των ICOs ή όχι, αρχικές προσφορές ICO και στα πλαίσια του κανονισμού θα πρέπει να μπουν τα ICOs, τα νέα νομίσματα έχει ξεκινήσει αυτή η αγορά και είναι θεμελιώδες ήδη να έχουμε ευρωπαϊκό regulation σε αυτό το πλαίσιο. Υποστηρίζω λοιπόν τη θέση του εισηγητού όπως υποστηρίζω και τη θέση του εισηγητού για τη ρύθμιση που δεν πρέπει να επικεντρώνει την εποπτεία στην ΕΣΜΑ. Είναι σημαντικό αντιθέτως να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών αρχών δοθέντως ότι έχουν μεγαλύτερη τεχνογνωσία και εμπειρία των εθνικών συστημάτων. Και δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ένας κανονισμός αυτού του είδους εφαρμόζεται με ρυθμίσεις σε επίπεδο εθνικό, όπως το προσπέκτους, ε, το MIFID και το σύστημα βαθμολόγησης για την ισοδυναμία για τρίτες χώρες. Ο εισηγητής σπρώχνει, θέλει να βάλουμε και τρίτες χώρες σε, αυτή, σε αυτές τις διατάξεις. Κατά την άποψή μου, συνδέεται η κατάσταση με το Brexit και είναι αρκετά προβληματική η κατάσταση και πιστεύω ότι για την ώρα θα πρέπει να παραμείνουν εκτός, να προβλέψουμε ίσως μια ρήτρα αναθεωρήσεως και ίσως αυτό θα ήταν καλό συμβιβασμό. Σε ένα, δύο χρόνια μπορούμε να το ξαναξετάσουμε για να ξέρουμε και τι θα μπορέσουμε να κάνουμε τις ζήτες χώρες. Όπως είπα, η ανταλλαγή απόψεων υπήρξε χρησιμότατη με τους συναδέλφους και σύντομα πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε λύσεις και τα τρία σημεία που παραμένουν ακόμα, κατά την άποψή μου, ανεπίλητα. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ, Μάρκο. Νομίζω κλείσαμε με τους σκιώδεις. Μίλησαν όλοι. Οπότε, ε, Περβάσου Πέρες. Ήθελα να πω δύο λόγια για δύο σημεία. Ο εισηγητής αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχαμε χθε με τους επικεφαλής των τριών εποπτικών ερχών. Μίλησαμε και για το συγκεκριμένο φάκελο, ούτως ή άλλως, εκ των πραγμάτων. Ε, και σημειώνω ότι ειδικά για τις αρχές προσφορές νομισμάτων, τα ICO, ο πρόεδρος της ΕΣΜΑ το είπε ευθέω. Πρόκειται για σοβαρό θέμα, απαιτητικό. Δεν είπαμε ποτέ όχι στην ε, καινοτομία, αλλά υπάρχουν κίνδυνοι ξεπλήματος, για παράδειγμα, χρήματος ε, υπό το κάλυμα της ανωνυμίας. Λέω στους συντονιστές ότι η καλύτερη λύση για την Επιτροπή μας θα ήταν την υπόθεση αυτή των ICO να την αντιμετωπίσουμε αλλά με τρόπο αυτό συνεπή. Δηλαδή να ξεκινήσουμε μια προφορική ερώτηση στην Κομισιόν με ή χωρί ψήφισμα και αυτό θα μας επιτρέψει πιστεύω να δώσουμε την ε, πρέπουσα σημασία στο θέμα. Όχι λοιπόν κάτι από σπόντα ή ε, παρόδο. Διότι το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν είναι δυνατόν να το αντιπαρέλθουμε έτσι με συνοπτικές διαδικασίες. Τώρα για το θέμα της ΕΣΜΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Άξιων και Αγορών, το θέμα των αρμοδιοτήτων της ε, ξανανοίγει. Ε, τι μπορεί να μας επαγορεύει να της προσδώσουμε μια επιπλέον αρμοδιότητα και μετά να δούμε ακριβώς πώς θα τα συντονίσουμε όλα αυτά. Βλέπω όμω μια αντίφαση αυτά που μας είπε ο εισηγητής όσον αφορά τις οδυναμίες ναι, δεν θέλουμε ένα διεθνές διαβατήριο για να φτιάξουμε μια τεράστια αγορά. Μας λέει εκεί είναι και μετά όταν έρχεται η ώρα της ρύθμισης αυτής της αρχής λέει α, όχι η νέα πλατφόρμα αλλά οι εθνικές αρχές. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι πρόκειται για μια μικρή αντίφαση εκτός αν δεν κατάλαβα καλά. Η πρόταση της Κομισιόν προκειμένου μου φαίνεται όσον αφορά δηλαδή, τον ρόλο της ΕΣΜΑ για να λειτουργήσει μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά είναι η καλύτερη πρόταση. Όπως άλλωστε το είπε και ο σκιώδης μας ε, και η κυρία Καηλή. Εντάξει, να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλήσει πριν ξαναμιλήσει ο Άσλε. Υπάρχει κάποιο από την Κομισιόν. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον συγγετή και του Σκιώδη ε, που εξέτασαν το κείμενο. Χαιρόμαστε που επετεύθη ταχεία πρόοδος, διότι είναι σημαντική πτυχία της ε, ενίας αγοράς κεφαλαίων και του σχετικού σχεδίου δράσεως για να χρηματοδοτούνται ναφείς επιχειρήσεις και διάφορες επιχειρήσεις. Τα τρία σημεία που συζητούνται στην Επιτροπή, ο ρόλος της ΕΣΜΑ, τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Ισότιμες συνθήκες, όρους ανταγωνισμού. Να μειώσουμε επίσης το βάρος επιπλατφορμών για να μπορούν να επιχειρούν στην ενή αγορά. Γι' αυτό υποβάλαμε κάποια πρόταση για να ζητήσουμε εποπτεία και αδειοδότηση των πλατφορμών μέσω της ΕΣΜΑ. Κατά την άποψή μας, συνάδει αυτό με το πνεύμα του να έχουμε συνεπείς κανόνες που ισχύουν για όλη την αγορά. Δεύτερον, για τα νέα νομίσματα, ICOs, ρητά δεν συμπεριλάβαμε τα νομίσματα αυτά στην πρότασή μας, γιατί, διότι χρειάζεται να μελετήσουμε και να αξιολογήσουμε το πώς αυτή η αγορά εξελίσσεται, ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν και πώς μπορεί να καλευθούν σε εποπτικό επίπεδο. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πρόημο αυτά τα καινούργια νομίσματα να τα, να τα συμπεριλάβουμε στην πρόταση αυτά κάθε αυτά. Προτιμούμε να ολοκληρώσουμε τις αξιολογήσεις μας και να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς στα μέτρα του τομέα για την ισοδυναμία τρίτων χωρών. Δεν συμπεριλάβουμε κάτι τέτοιο στην πρότασή μας, διότι οι αγορές στην Ευρώπη έχουν πολύ μικρό ποσοστό πληθοπορισμού, κυρίως εν συγκρίση με άλλες περιοχές όπου είναι η Ασία και οι Ηνωμένε Πολιτείες. Σκοπό τη προτάσεως είναι να αυξηθεί η αγορά και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την ενιαία αγορά, ούτω ώστε αυτέ οι πλατφόρμες να αναπτυχθούν σε όλη την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Καλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν συνοψίσει ο Άσλε να πω κι εγώ κάτι. Και εγώ έχω αποβάλει σχετικέ τροπολογίες. Καταρχά ευρεία συμφωνία όσον αφορά το όριο, πιστεύω. Αυτό διευκολύνει τα πράγματα και για τους σκιώδεις και για τον εισηγητή, για την ισοδυναμία. Τι είναι σαφές από την έκθεσή μας που ετοιμάσαμε εδώ και κάποιος μήνες θετήθηκε από το Κοινοβούλιο. Η Γενική Αρχή μας βρίσκει συμφώνους. Όταν μια χώρα συμμορφώνονται με το ρυθμιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα καθοριστέντα πρότυπα και τις ενδεδειγμένες νομικές διακρίσεις που προβλέπονται, Καταρχή, αυτή η τρίτη χώρα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί στην αγορά μας. Το επιχείρημα που αναφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια λιγότερο ανεπτυγμένη αγορά αναγνωρίζεται. Για να αναπτυχθεί η αγορά μας στο μέλλον πρέπει να ανοίξει, να ανοιχτεί σε τρίτες χώρες. Τρίτες χώρες που σαφώς συμμορφώνονται πλήρως με το ρυθμιστικό και υποπτικό μας σύστημα. Κάποια ιδέα άκουσα αναφέρθηκε η δυνατότητα αναθεώρηση του τομέα, ίσως να είναι κάτι ενδιαφέρον. Μπορεί να το εξετάσουμε περαιτέρω. Πολλά από αυτά τα θέματα ε, χάνονται στην πολιτική κατάσημερινή. σημερινή. Στην έκθεσή μα είπαμε ότι θα πρέπει αυτό να επεκταθεί και νομίζω αυτή είναι βασική αρχή. Για το θέμα το έσμα μέσω έναντι εθνικών αρχών είναι ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε σε, διπλό, σε καθεστώς διπλής αδειοδότησης. Δεν θα ήταν καλό αυτό για τις συναδειόμενες αγορές ούτε για τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες που δημιουργούνται. Ενδιαφέρουσα ιδέα που αναφέρθηκε, μιας νομικής γνωμοδοτήσης, ώστε να ξέρω ποια είναι η άποψη του Άσλι. Και χτες αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της ΕΣΜΑ ήταν ενδιαφέρον και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε κατά τις διαπραγματεύσεις. Ο Άσλι λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, σκιώδεις για τα σχόλιά τους. Δεν θα επαναλάβω τα σχόλια εφόσον μάλιστα θα διεξαχθεί το απόγευμα συνεδρίαση σκιωδών. Να απαντήσω σε ένα-δύο σημεία που εθίγησαν. Ευχαριστώ σας για τα σχόλια για την προστασία των επενδυτών. Υποβάλλατε και σχετικές τροπολογίες, τις έχω λάβει υπόψη. Λοιπόν, και μέσω των ε, δοκιμών ε, περιγνώσεων ε, μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτήν την ιδέα. Θέλω να εξετάσω την ιδέα σας περί νομικής νομοδοτήσεως. Τι πρόβλημα έχω, ίσως έτσι καθυστερήσει κατά πολύ η όλη διαδικασία. Δεν θα πω ναι ή όχι τώρα. Θέλω να το σκεφτώ. Μόλι αναφέρθηκε σε δύο τροπολογίε, στην 249 και 282, να τι εξετάσω. Κυρίως αυτή που αναφερόταν στις κεφαλοχικέ απαιτήσει και τη σχετική τροπολογία. Εύα και Μάρκο, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, για τα νέα αυτά νομίσματα, τα ICOs. Υποψιάζομαι ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το ψηφίσουμε στην ε, Επιτροπή. Ε, εκεί δεν έχουμε κοινή άποψη, ισκιώδης, και φαντάζομαι ότι οι δύο μεγαλύτερες ομάδες έχουν διχασμένες απόψεις. Είναι διχασμένες και οι δύο ομάδες. Και για να λυθεί το θέμα είναι να ψηφίσουμε. Ε, δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου. Ίσως να είναι εντελώς αντίθετο. Εν τη αυτή περιπτώσει τελειώνει ο χρόνος και θα τα βγάλουμε πέρα. Εμείς σαν Κοινοβούλιο θέλουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται και θα πετύχουμε και περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ψηφίσουμε και αν συμπεριλάβουμε την προσέγγιση μας στο κείμενο. Προτείνω λοιπόν να ε, περιλάβουμε, συμπεριλάβουμε τα νέα νομίσματα Εσύ ως Εύα αναφέρθηκε σε ισοδυναμία και ίσως ότι θα χρειαζόταν μια αναθεώρηση στο μέλλον επ' αυτού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε προσεκτικά συντάσσοντας τις συμβαστικές. Πρόεδρε, εδώ είναι τα τελειώντα σχόλιά μου και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Άσλη. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόγραμμα. διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ψηφοφορία στην Ίκον 5 Νοεμβρίου. Καλή τύχη στους Σκιώδης και στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Δύο λεπτά διάλειμμα και θα ξαναρχίσουμε όταν είναι εδώ και ο Ζουροζάτη. So, thank you, colleagues. Λοιπόν, ευχαριστώ συνάδελφοι. Πάμε στο σημείο 14 και 15 στη μέση διάταξη. Οι κανόνες που συνδέονται με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων σε μια σημαντική ψηφιακή παρουσία. Και το 15 κοινό σύστημα ε, για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ε, τα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών. Πρώτο θέμα λοιπόν, φορολόγηση των εταιριών με σημαντική ψηφιακή παρουσίαση. Γιατί είναι ο κύριο Ντάριο Ροσάτη αλλά ο κύριος Λούντβιχ θα πάρει το λόγο εξ ονόματος του εισηγητού. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Με χαρά αντικαθιστώ το συνάδελφο και φίλο ε, Ντάριους Ροσάτη. Ε, ζητεί συγγνώμη για την απουσία του. Θα σας διαβάσω επιλέξει ε, τη δήλωσή του για αυτό το σημαντικό θέμα. Και πάλι ο Ντάριους θα ήθελε να τονίσει ότι υποστηρίζει τη γραμμή της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκθεση αυτή. Θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντική στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται στον ΩΣΑ για την ψηφιακή οικονομία. Και μάλιστα δεν επιβάλλεται επιπλέον φόρος. Στον ΩΣΑ πρέπει να γίνει λοιπόν η συζήτηση και η συνεννόηση σε αυτό το πλαίσιο. Καλωσορίζουμε την προσπάθεια αυτή, αλλά δεν έχει ακόμα προχωρήσει αρκετά. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει να προχωρήσει. Τονίζει παρόλα αυτά ο Ντάριο ότι η οδηγία αυτή θα πρέπει να αποτελεί στη βάση για περαιτέρω συνεργασία σε διεθνέ επίπεδο. Επειδή δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση έχουν αρχίσει τα κράτη-μέλη να προχωρούν σε μονομερείς κινήσεις και αυτό σημαίνει κατακαιρματισμό της ε, ψηφιακής ενιαίας αγοράς και αβεβαιότητα. Αυτά θα πρέπει να αποφεύγονται. Πάντω, λέει ο Ροζάτη ότι δεν αλλάζει ουσιαστικά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή του. Ασχολείται με διάφορα σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, θα πρέπει να σημειώσουμε ε, ε, τι εργασίε των επιτροπών τάξε, τάξε 2 και πάνω ε, για την ψηφιακή οικονομία. Δεύτερον, τονίζει ο Ντάριο Ροζάτη ότι βάσει μάλλον λόγω της αβεβαιότητας ε, που συνδέεται με τον ορισμό, τι σημαίνει σημαντική ψηφιακή παρουσία και ε, ε, ψηφιακές υπηρεσίες. Θα πρέπει να υπάρξει σαφής ορισμός των δύο ενιών έτσι ώστε και οι εταιρείες αλλά και οι εφορίες να μειώσουν την αβεβαιότητα που επικρατεί. Έχουν τονίσει πολύ ενδιαφερόμενοι ότι είναι πρόβλημα ε, η έλλειψη ορισμών. Τονίζει επίσης ο Ντάρης ότι η Επιτροπή της Ψηφιακής Φορολογίας Ε, τονίζει ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά η οδηγία από τις εταιρείε. Οι εθνικές φορολογικές αρχές θα πρέπει να αξιολογούν ε, και να εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες και να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ ε, των άλλων φορολογικών αρχών, όλων των ευρωπαϊκών, για να μην υπάρχει διπλή φορολογία ή υπερφορολόγηση δεν προτείνει συγκεκριμένη δομή ο Ντάριος Ρωσάτη. Η έκθεσή του επίσης υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία θα πρέπει να σέβονται την αρχή της ουδετερότητας του φόρου και να μην κάνουν διακρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκές και μη εταιρείε. Ω προ το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Και τέλο, αλλά είναι και αυτό σημαντικό, προ το παρόν ο Ντάριος δεν θέλει να αλλάξει κανένα κατόφλι για το τι σημαίνει σημαντική ψηφιακή παρουσία. Χρειάζονται μελέτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του ενεχομένους για να γίνουν οποιασδήποτε αλλαγέ και όχι αυτά να γίνονται στην τύχη και κατά το δοκούν. Αυτά. Στη διάθεσή σας ο εισηγητής και σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λούτβιχ, εξ ονόματος του Τάριου Σροσάτη, παρουσίασε στην έκθεσή του. Και το επόμενο θέμα, κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών. Ο Πολ Τάγκ είναι η συγκητής μας, έχει το λόγο, στα αγγλικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Μπράιν. Σήμερα συζητάμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο και πληρώνουν τους χαμηλότερους φόρους. πολλοί το θεωρούν κάτι άδικο και εντελώ αναποτελεσματικό. Δεν είναι ισότιμη όρη επικρατών. Οι αριθμοί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ μεταξύ παραδοσιακών πολυεθνικών και ψηφιακών πολυεθνικών. Κυρίω όταν ψηφιακέ πολυαθνικέ κάνουν ένα πολύ επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Οι μεγαλύτερε εταιρείε στον κόσμο έχουν τη χαμηλότερη φορολόγηση. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Τούτων λεχθέντων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη στις εκθέσεις Αλέν Λαμασούρ και στη δική μου για το CCTB και το CCCTB προτείνουμε διαθετικές λύσεις. Στο τέλος πρέπει οι εταιρείε να πληρώσουν μεγαλύτερο εταιρικό φόρο, φόρο επί των κερδών και σε αυτές τις εκθέσεις έχουμε την έννοια της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας. Ευπρόσδεκτη συζήτηση από αυτού του θέματος. Ταυτοχρόνως γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο κινείται αργά, ούτως υπήν. Και το Συμβούλιο θα πρέπει να κινηθεί πέραν της ομοφωνίας, να κινηθεί προς την πλειοψηφία στις ψηφοφορίες για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Είναι τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Χρειαζόμαστε και σύντομα, ε, βαχυπρόθεσμα κάποια λύση. Και να μην μπλοκάρουμε τις αναγκαίες διαθροτικές λύσεις. Χαίρομαι, διότι και οι Γάλλοι έχουν υποβάλει με ρήτρα σταδιακής κατάργησης, δείχνοντας ότι όλη η ρύθμιση είναι προσωρινή. το στηρίζω αυτό. Από βραχυπρόθεσμα θέλουμε να κινηθούμε προς το μακροπρόθεσμο, να βρούμε μια μακροπρόθεσμη διαθροτική λύση. Συζητήσαμε, άμα συζητήσουμε τη βραχυπρόθεσμη λύση, δεν υπάρχει λόγος να μην επιδιώξουμε ισότιμους όρους για όλους. Τι πιστεύω. Ότι τώρα το ποσοστό φορολόγηση 3% είναι πολύ χαμηλό, συντελεστής πρέπει να είναι κοντά στο 5% λόγω των περιθωρίων κέρδους που υπάρχουν. Κυρίως όταν γίνεται ένας επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός, 3% είναι χαμηλό, 5% είναι καλό, δεν θα πρέπει να εξαιρέσουμε τις μεγάλε εταιρείε και τις αυξανόμενες, τις, αυτές που αυξάνονται σε μέγεθος. Η Emerson είναι από τις μεγάλε εταιρείε στον κόσμο. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση για τις πλατφόρμες, για τις ψηφιακές εταιρείε. Να αυξήσουμε και το συντελεστή και το πεδίο εφαρμογή και να, να συμπεριλαμβάνουμε και την Emerson και την Netflix. Να είμαστε πιο φιλόδοξοι πρέπει. Και το σωστό μήνυμα πρέπει να φύγει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν βρίσκει τη λύση το Συμβούλιο. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι χρειάζεται δράση. Φιλόδοξη δράση. Και θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι στο μέλλον από ό,τι τώρα. Να στείλουμε σωστό πολιτικό μήνυμα ότι χρειάζεται πρόοδος. Μεγαλύτερη κάλυψη, υψηλότερος φορολογικός συντελεστής. Και θα πρέπει να συζητήσουμε και τη σημαντική ψηφιακή παρουσία. Υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί της ψηφιακής παρουσίας. Στο CCTB ορισμός είναι ευρύτερος από ότι αυτός που υιοθετήθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να το συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο. Τέλος, να συμπληρώσω κάτι. Ποια είναι η κατάσταση. Οι εθνικές φορολογικές αρχές θα ασχοληθούν με ευρωπαϊκούς φόρους. Προς τα εκεί πάμε. Πρέπει να δούμε και τα πρακτικά ζητήματα. Οι εθνικές φορολογικές αρχές πώς τα καταφέρνουν. Ίσως χρειάζεται έλεγχος. Έλεγχος ομοτήμων όσον αφορά τις εθνικές φορολογικές αρχές. Πώς ασχολούνται με το DST, διότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Ότι κάθε φορέας που ασχολείται με αυτά τα θέματα, με τους ευρωπαϊκούς φόρους, ασχολείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πολ. Οι δύο σύντες μίλησαν από το... Δηλαδή, ΕΛΚ και σοσιαλιστές μίλησαν από ECR. Ο κ. Φόξ είναι ο Σκιώδης, αλλά νομίζω ο Μπέρναρτ θέλει να μιλήσει και θα μιλήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Ασουλέη ζητά συγγνώμη, κολλείεται και μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόματός του. Για την Επιτροπή Ροζάτη. Ο εισηγητής υπέβαλε δύο τροπολογίες επί του σχεδίου. Ας λέει, συμφωνεί με την φορολόγηση αυτών των εταιριών. Είμαστε υπέρ των τροπολογιών του εισηγητή με τις οποίες υποστηρίζεται η δουλειά του ΩΣΑ του θέματος με προστασία όμως της κυριαρχίας των κρατών μελών στα θέματα εταιρικού φόρου. Καταλαβαίνει ότι τα 7 εκατομμύρια είναι το κατόφλι όμως ε, δεν ξέρω αν πρέπει αυτό να περιπληθεί στο CCCTB. Η ομάδα μου επίσης θεωρεί ότι ιδανικά τα μέτρα του ΩΣΑ πρέπει να εφαρμοστούν, αν και αυτό δεν φαίνεται πολύ πιθανό σε αυτή τη φάση. Οπότε τα κρατημέλη μεταξύ δεν πρέπει να εμποδιστούν να λαμβάνουν μονομερός μέτρα ο κύριος ε, Φόξ θα συνεργαστεί ευχαριστώ φυσικά με τον ΣΥΤΗ για το θέμα και έχω και μια δεύτερη δήλωση εδώ του κυρίου Φόξ για την Επιτροπή για την έκθεση με και πάλι συμφωνεί γενικά με το κείμενο, συμφωνεί με τη φορολόγηση της πώληση στοιχείων, δεδομένων, Ανισχύει όμω ε, με την επέκταση του αντικειμένου αυτής της έκθεσης Προτείνει επίσης μια αύξηση του ποστού σε 5% από 3% που προτείνει η Κομισιόν και υπογραμμίζει ότι είναι ένα ενδιάμεσο προσωρινό μέτρο εν CCCTB και προτείνει ρήτρα μετάβασης. Επίσης είναι κατά της επέκτασης του αντικειμένου του πεδίου εφαρμογή χωρίς μελέτη επιπτώσεων. Το θέμα είναι να γράψουμε κάτι το οποίο να έχει προσθεμένη αξία. Επίσης, ως ECR, ε, ε, και όπως είπα και για την έκθεση Ρωσάτη, δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε τα μονομερή μέτρα των κρατών μελών. Πιστεύω λοιπόν ότι τα μέτρα του πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά επειδή, όπως είπα, δεν θα γίνει αυτό μάλλον πολύ σύντομα, ε, δεν πρέπει να εμποδίσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν μόνο μέτρα. Αυτό ισχύει και τις δύο εκθέσεις, Ροζάτη και Τάν. Και βεβαίως είμαστε στη διάθεση του εισηγητή για συνεργασία. Πρόεδρος. Από την άλλη δεν είναι κανείς, από ό,τι βλέπω. Πράσινη. Είναι κανείς εδώ. Από την Κούα είναι ο Μάρτιν. Μάρτιν, αν θέλεις να μιλήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συζήτητες. Ε, πραγματικά έχουν δίκιο. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τα σχέδια των εκθέσεων τους. Τα θέματα αυτά μας απασχόλησαν και στην προηγούμενη συζήτηση και σήμερα και τώρα. Στον 21ο αιώνα το φορολογικό ε, δίκαιο θα πρέπει να αφορά ε, και τις εξέλιξεις κοινωνίας και την ψηφιακή οικονομία που θα πρέπει να πληρώνει το μερίδιο του φόρου που της αναλογεί. Πολύ ενδιαφέρον θέμα και για μας de facto είναι πώς θα συμμετέχει στην αναδιανομή του πλούτου, ο πλούτος που έχει παραχθεί και ε, στην ψηφιακή οικονομία. Έχουμε διάφορα φορολογικά σκάνδαλα, τα οποία ακούσαμε προηγουμένως, εταιρείε ε, του διαδικτύου και μεγάλη ψηφιακή ε, όμιλη και κολοσσή δυστυχώς ήρθαν αρνητικά στη δημοσιότητα. Και η θέση του νομοθέτη, αν μου επιτρέπουν οι συνάδελφοι, στο παρελθόν αξίζει μια μεταφορά έτσι, ε, αγγλοσαξονικής κοπής που είναι οι δύο ηλικιωμένοι στο Muppet Show που το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να σαρκάζουν και να σχολιάζουν ηρωνικά τα όσα συμβαίνουν επί σκηνής. Λοιπόν, επειδή είμαστε αυτοί εμεί στη ε- ε- ε- Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό είναι να φύγουμε από το θεωρείο και να πάμε στη σκηνή και να είμαστε και πρωταγωνιστέ σε αυτή τη ψηφιακή οικονομία και να πληρώσει το μερίδιο των φόρων που τη αναλογεί η ψηφιακή οικονομία. Δυστυχώ εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τι τελευταίε εβδομάδε ακούμε πολλέ επικριτικέ φωνέ από διάφορα κράτη-μέλη ω προ την εισαγωγή ενό φόρου των ψηφιακών υπηρεσιών. Και μάλιστα η γερμανική κυβέρνηση είναι πάρα πολύ επιφυλακτική. Διαφωνώ ρητά και ελπίζω και ο Γερμανός Υπουργό Οικονομικών να αλλάξει τη θέση του, να αναθεωρήσει. Και βεβαίως χρειάζεται ψηφιακός φόρος που θα σε διαμορφώσουμε και εμεί. τώρα για τη συγκεκριμένη έκθεση, τις δύο εκθέσει καλύτερα. Για μας η αρχή είναι ότι φορολογεί όπου ε, έχεις οικονομική δραστηριότητα και κέρδη. Ε, ο κύριος Ροζάτη που δεν ξέρει πώς θα ορίσει την ψηφιακή παρουσία ε, θα ήθελα να μου απαντήσει γιατί δεν το έχω καταλάβει στην επόμενη συζήτηση για την έκθεση για ποιο λόγο είναι τόσο πολλές εξαιρέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλω να υπερφορολογούνται προφανώς αλλά εάν ξεχυλώσει τόσο πολύ το θέμα των εξαιρέσεων, θα έχουμε ένα παράλληλο φορολογικό σύστημα που δεν είναι καθόλου σκόπιμο Και σε σχέση με την τροπολογία νέα θέλω κάτι να ρωτήσω που γίνεται σωστά αναφορά ε, στις αρμοδιότητες των κρατών μελών στα φορολογικά. Αλλά αυτό βλέπω να είναι σε κάποια αντίφαση με την έκθεση ΤΑΝΚ. Εμεί, ω νομοθέτη, μπορούμε να ορίσουμε ένα φορολογικό συντελεστή για να μην υπάρχει κούρσα προς τα κάτω γιατί υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι αν εγκριθεί η τροπολογία 9. Ναι. Έρχομαι τώρα στην έκθεση ΤΑΝΚ. Ε, χαιρόμαστε για την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο 5%. Το υποστηρίζουμε και εμείς και θέλουμε να διευρυνθεί και το ε, πεδίο εφαρμογή και σε άλλες πλατφόρμες για να μπορέσει η ψηφιακή οικονομία να συνεισφέρει και να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στην κοινωνία θα συνεργαστούμε επικοδομητικά και για τις δύο εκθέσεις και ελπίζουμε να είναι αρκετά χειρό το μήνυμα που θα στείλουμε από κοινού στο Συμβούλιο για να αλλάξουν γνώμη και οι επιφυλακτικοί και οι σκεπτικιστές στα διάφορα κράτη-μέλη και ο Γερμανός υπουργό Οικονομικών. Ευχαριστώ Μάρτιν. Η FTD. Επόμενη ομάδα, αν είναι κάποιος εδώ. Παρακαλώ, όχι, όχι. Από την ΕΝΕΦ. E Ούτε. Οπότε, ποιο θέλει να μιλήσει. Α, άλλον δεν σε είδα, συγγνώμη. Πρόεδρε, συγχαρητήρια στον εισηγητή, εξαιρετική εργασία. Το κείμενο είναι μια πολύ καλή βάση εξαίρεση του θέματος για την Επιτροπή μας. Το έκαναν και άλλοι. Θέλω να επιμείνω στον κατεπήγοντα χαρακτήρα της έκθεσης. Το είπαν και άλλοι. Γιατί, διότι κάποια κρατημέλη, από τι φαίνεται υπό την πίεση της κοινή γνώμης, αλλά και για άλλους λόγους, ε, είναι έτοιμα να λάβουν μονομερείς αποφάσεις, κάτι το οποίο είναι παραλόγω σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, ελπίζω ότι ακόμη δεν έχουμε χάσει την ευκαιρία και μετά από τα διάφορα σκάνδαλα φοροποφυγής, ε, απόκρυψη φορολογικού εισοδήματος, μεταφοράς κερδών από τις εταιρείε. και ότι κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν ε, και από εμά και από την Επιτροπή, την Κομισιόν, όπως είπα για να αξιοποιήσουμε αυτά τα σκάνδαλα έτσι ώστε να θεσπίσουμε ένα σύστημα φορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αν γίνεται, το οποίο θα είναι πιο ικανοποιητικό σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση. Προσθέτω συναφώς ότι ω πρόσφατα οι πρωτοβουλίε που θα μπορούσε, θα μπορούσε να, να έχει λάβει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίφθησαν ως απειλές ε, κατά το καλύτερο κομματιού της αμερικανικής οικονομίας μέσω δηλαδή αυτών των φορολογικών μέτρων. Χάρη σε, αυτή τις, αυτές κάποιες ε, εταιρείε κάτσαν στο σκαμνί, το σπιν και αυτό θέλαμε όπως κάνουμε και με την προστασία των ε, δεδομένων. Το επιχείρημα ορισμένων τώρα είναι το εξή. Ο ΩΣΑ κάνει τη δουλειά του. Περιμένουμε τον ΩΣΑ. Είναι λεπτό το θέμα. Α περιμένουμε. Μα δεν περιμένουμε. Οι Αμερικανοί δεν περίμεναν τον ΩΣΑ για να μεταρρυθμίσουν εκ βάθρων το φορολογικό του σύστημα και δει την αντιμετώπιση των πολυεθνικών, των Αμερικανικών πολυεθνικών και των θηγατρικών τους ή των θηγατρικών των Ευρωπαϊκών πολυεθνικών. Λοιπόν, έχουμε ένα στόχο. Ξέρουμε τι θέλουμε, α το κάνουμε. Να παρακολουθούμε φυσικά παράλληλα το έργο το οποίο γίνεται στον ΩΣΑ. Φυσικά να είμαστε σε συνεννόηση με τους εταίρους μα στον ΩΣΑ, έστω και στο περιθώριο του ΩΣΑ, αλλά, αλλά δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει ε, προπετούμενο η ολοκλήρωση του έργου στον ΩΣΑ. Τώρα στους νέους ιδίου πόρου, χάρη στου οποίου θα πρεκοδοτήσουμε τον προπολισμό μα. Η Κομισιόν προτείνει και μια ενοποιημένη φορολογική βάση για τα τερικά κέρδη. Αυτό το συζήτησαμε χθε. Αυτό δίνει στην πρόταση τη Κομισιόν έναν μάλλον οτοπικό χαρακτήρα στην πρόταση αυτή. Δεν ζούμε σε ένα ιδιαίτερο κόσμο, τον οποίο θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε μέρο του προπολογισμού, του ενωσιακού προπολογισμού με φορετεριών. Εδώ θυμίζω απαιτείται ομοφωνία ενώπιση του επομένου π. Άρα λοιπόν όλα αυτά κρατήρουν στο ότι είναι κατεπήγον το θέμα και για εμάς εδώ αλλά και στο Συμβούλιο. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν, η οποία εκπροσωπείται διόνως εδώ. Ε, η Κομισιόν πώς βλέπει το θέμα, πού πηγαίνουμε από εδώ και πέρα και πού θα πάμε στο Συμβούλιο. Και κλείνω λέγοντας ότι αν, είναι, αν υπάρχει ένα θέμα επί του οποίου μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε, ε, εκεί πρέπει να συμφωνήσουμε το Κοινοβούλιο και τα λαθισμικά όργανα, είναι η φορολόγηση της ψηφιακής παρουσίας. Αυτό λέει και ο Τάγκ, λίγο πολύ, και ο Ροζάτη. Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να ορίσουμε και την ψηφιακή παρουσία. Με τον Τάγκ το είδαμε στην έκθεση την ενοποιημένη φορολογική βάση και τη εταιρεία. Εντάξει, θα το δούμε, το βελτιώσουμε, αλλά ε, νομίζω ότι αν είναι κάτι να κάνουμε, αυτό είναι το θέμα που πρέπει να μα απασχολήσει και να, από αυτού πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ, αλλά κάποιος από τους ομιλητέ μας κατέφθασε. Η κυρία Φοντινέ Λόπε του ΕΛΚ. Αν έχετε συγκεντρωθεί, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο που θέλω να πω, Πρόεδρε, είναι να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για τις προτάσεις που έχουν κάνει και το έργο τους ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του κυρίου Μάτο που κολλείεται και δεν μπορεί να είναι παρόν γιατί έχει ψηφοφορίες στο ΕΛΚ, στο Επιτροπή Αλίας, συγγνώμη, που είναι συντονιστής του ΕΛΚ. Έχουμε ταυτόχρονα πολλές ψηφοφορίες σήμερα. Ε, η ε, ενιαία ψηφιακή ε, αγορά θα πρέπει να είναι πολιτική προτεραιότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Χρειάζεται να σχεδιαστεί ένα σύγχρονο και σταθερό φορολογικό σύστημα για να ανοίξουν ψηφιακές δυνατότητες για πρόσωπα και εταιρείε σε μια αγορά ε, τη ευρωπαϊκή Ένωση με πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Συμφωνώ με τον κύριο Τάνγκ ότι είναι ένα προσωρινό μέτρο αυτό μέχρι, για να λυθεί κατεπηγόντως η κατάσταση έτσι ώστε όλες οι επιχειρήσεις να πληρώνουν τη φορολογία που τους αναλογεί και να συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή οικονομία και να υπάρχει και θεμητός ανταγωνισμός για τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Ο κύριος Μάτο θεωρεί ότι κάθε εταιρεία θα πρέπει να πληρώνει το φόρο που της αναλογεί όπου της αναλογεί. Εκτός αυτού και εκτός της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής και τα φορολογητέα κέντρη και οι ψηφιακές υπηρεσίες που μπορεί να είναι οπτικοακουστικές ή κείμενο και επιγραμμικές μέσω ε, ψηφιακών πλατφορμών. Η πρόταση που μας έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και πρωτοπόρα και φιλόδοξη, αλλά υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα φορολογητέα κέρδη ε, με μελέτη αντικτύπου και μάλιστα λεπτομερή και εμπεριστατωμένη. Και δεν είναι μόνο αυτό, θα πρέπει να προχωρήσουν οι συζητήσει και οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο, γιατί κινδυνεύουμε εκεί πολλά κρατημέλη να αποφασίσουν ε, να προχωρήσουν στις δικές τους ε, προτάσεις παραβιάζοντας έτσι την εσωτερική αγορά. Θέλησε να τονίσει δύο βασικά σημεία κύριος Μάτο. Πρώτον, την ανάγκη να υπάρχει μια εποπτική αρχή που θα ε, εποπτεύει πραγματικά την, την ε, ίσπραξη αυτών των ε, φόρων όπου οφείλουν να καταβάλουν το φόρο οι εταιρείε και να υπάρχει μια αυστηρή ρήτρα αναθεώρησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων αυτών των μέτρων και αν χρειαστεί να συμπεριληφθούν και άλλες υπηρεσίες στο πεδίο εφαρμογή. Αυτά και τίποτα άλλο και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε κάποιες ερωτήσεις και άκουσε παρατηρήσεις. Θέλει να πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλει, υπάρχει ευκαιρία να μιλήσει. Ε, bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Καλημέρα, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τον εισηγητή διεξοδικότατη ανάλυση των προτάσεων που κάναμε για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Στην έκθεση TONG το θέμα που αφορά το πεδίο εφαρμογή διασυνδέει το βραχυπρόθεσμο με το αποκρόθεσμο. Πολύ καλό αυτό. Είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ξέρετε ποιε είναι οι προτάσει μας. Είμαστε βεβαίω στη διάθεσή σας. Μπορούμε να σας δώσουμε την τεχνογνωσία μας όσον αφορά τα πιο καινούργια στοιχεία που εντοπίσατε. Στην έκθεση του κυρίου Ροζάτη αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι η σχέση με τις εργασίες αυτής, τη της Επιτροπής όσον αφορά την ενιαία φορολογική βάση των εταιριών. Είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να συζητείται στο Συμβούλιο. Οι φόβοι που εξεφράστησαν για το ψηφιακό πακέτο και ότι αυτό θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή από τι εργασίε του STB, θέλουμε να μην είναι κάτι που θα υλοποιηθεί. Και ο συσχετισμό μεταξύ των δύο θα πρέπει να εξακολουθεί να εξετάζεται. Ο κ. Λαμασούρ ρώτησε αν μπορούμε να ενημερώσουμε για τις συζητήσεις στο Συμβούλιο. Να περιοριστώ στις τεχνικής φύσεως ε, συζητήσεις πολιτικές παρακολουθείτε όπως και εμείς από τον τύπο και τις θέσεις των διαφόρων υπουργών. Τεχνικός πώς. Η Ευστρική Προεδρία έκανε εξαιρετική δουλειά σταθεροποίησης του κειμένου. Τα σημεία που σε επίπεδο τεχνικό εξακολουθούν να συζητούνται δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα. Αφορούν το πεδίο εφαρμογή, όπως γνωρίζετε, αντίθετα από αυτά που ο κύριος Τόγκ προτείνει, το Συμβούλιο προσπαθεί να μειώσει το πεδίο εφαρμογή σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, κυρίω όσον αφορά το θέμα των πωλήσεων στοιχείων. Άλλο θέμα που συζητείται αφορά τη ρήτρα σταδιακή εξάλληψη, τη ρήτρα αναθεώρησης. Όπως ο Υπουργό Λεμέρ ανακοίνωσε, είναι επιτάπητο των συζητήσεων του Συμβουλίου, προσπαθούν να βρουν ένα κατάλληλο κείμενο, μια διατύπωση αποδεκτή. Τρίτο σημείο, αυτό αφορά τη συζήτηση επί της συλλογή του φόρου, εις πράξεως του φόρου, ούτως ώστε το διοικητικό άχθος για τα κράτη-μέλη να μην αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτά είναι τα τρία σημεία που συζητούνται. Η Αυστριακή Προεδρία ελπίζει γρήγορα να πετύχει συμφωνία και έτσι η πολιτική σφίσο συζήτηση να στηριχθεί επικειμένου τελικού που θα αποφασιστεί σε τεχνικό επίπεδο. Όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάθεση του εισηγητού και των σκιωδών για κάθε τεχνική φύσεως ερώτημα που θέλουν να απαντηθεί και να επενθυμίσουν την πλευρά μα, όπω και σήμερα το πρωί, ότι είναι κατεπίγουσα η ανάγκη λήψεω αποφάσεω επ' αυτού του θέματο. Διότι τα κράτη-μέλη, όπω παρουσιάζουν τον προπολογισμό του για το καινούριο χρόνο, βλέπουμε πολλαπλασιασμό των φόρων που αποφασίζουν αυτά τα κράτη-μέλη. Άρα δεν είναι αν θέλουμε ψηφιακή, φορολόγηση ψηφιακών υπηρεσιών ή όχι, αλλά ποιο θα είναι ότι θα είναι δύσκολο να έχουν πολλού φορολογικού συντελεστέ και να υπάρξει ε, Συντονισμό αν υπάρχουν τόσοι πολλοί φορολογικοί συντελεστές διαφορετικοί του χρόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλο συνάδελφος που θέλει να μιλήσει. Έχω και εγώ κάποια σχόλια. Καταλαβαίνω. Δύσκολο το ζήτημα. Δύο θέματα έχουμε. Το πραγματικό πρόβλημα. Τι κάνεις με τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας σήμερα υπό τις παρούσες περιστάσεις. Έχεις μεγάλη ποικιλία επιχειρηματικών μοντέλων. Πνευματικά δικαιώματα, διανομή, διάθεση στην αγορά, παρασκευή, παραγωγή. Ε, δύσκολο όλα αυτά να καλυφθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον. Άλλο πρόβλημα, πολιτικής φύσεως. Υπάρχει αίτημα του κοινού για ασφάλεια φορολόγηση σε αυτό το τομέα. Να υπάρχει φορολόγηση. Όπω ξέρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 8-9% είναι ο φορολογικό συντελεστή, ο μέσο όρο. Πολύ πιο χαμηλά από ό,τι για άλλε εταιρείε, μεγάλε και μικρέ, που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ο συντελεστή του τομέα πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπω αναγνωρίζει στην έκθεση ε, Ροζάτιο, το θέμα τη κυριαρχία για τη φορολόγηση. Επίσης, ο Αλένα Μασούρ έθεσε το πρόβλημα. Πώς προσπαθούμε να πετύχουμε συνένεση. Καλύτερα να το κάνουμε αυτό βασιζόμενοι επί συμφωνίας, παρά μέσω μονομερών θέσεων που μπορεί να στρεβλώσουν την ενιαία αγορά. Αυτό κυρίως στον τομέα τον ψηφιακό. Διότι αν υπάρχει τέτοια διεθνοποίηση, είναι τόσο διεθνή, διεθνής ο χαρακτήρας αυτής της αγοράς και τέτοια μεγάλη ποικιλομορφία. πρόθεσμα είναι διεθνή συμφωνία στο μοντέλο του ΟΣΑ, πιστεύω. Παραμένει όμως το θέμα αυτό πώς εφαρμόζεται όταν βλέπουμε ότι οι ακολουθούν σαφώς διαφορετική κατεύθυνση. Ο ΩΣΑ είναι ανοιχτό, Έχει παράξει ένα έργο που δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα εξέβρεση λύσεως. Ο Επίτροπος Μοσκοβίτς είχε πει κάτι την περασμένη φορά. Μπορούμε να δούμε μήπως μπορούμε να έχουμε μια πρόταση με ρήτρα σταδιακής εξάλληψης, σταδιακής κατάργησης. Ίσως στα πλαίσια του BEPS ε του ΟΣΑ να βάλουμε τη φορολόγηση ψηφιακών υπηρεσιών και ίσως έτσι να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το τέλμα. Ίσως τα κράτη-μέλη πρέπει να το δουν αυτό. Εάν τα όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη θέλουν να δουν πώς στη δική τους δικαιοδοσία θα φορολογήσουν τις ψηφιακές ε, υπηρεσίες και πώς θα ενταχθεί αυτό στον προϋπολογισμό τους. Υπάρχει μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι, αλλά αυτό πρέπει να γίνει επί τη βάση συνένεσης. Τι σημαίνει αυτό, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να υποχρεωθούν να κάνουν κάτι όταν θεωρούν ότι θα χάσουν κάτι. Στο μηχανισμό αποζημίωσης και προς μια διεθνή συμφωνία, στην πορεία προς διεθνή συμφωνία, ίσως μπορούμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε. Αυτές είναι οι σκέψεις που έχω. Αν Ρούντι και ο Πολ θέλουν να πούν κάτι. Ο Πολ έχει να πει κάτι. Ορίστε Πολ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι υπάρχει ζήτηση του κοινού, όπως την αποκαλέσατε, για δίκαιη φορολόγηση και ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Πράγματι, ποιο είναι ο κίνδυνο. Αν δεν συμφωνήσουμε στην Ευρώπη, θα ακολουθηθεί μονομερής προσέγγιση και κατακαιρματισμός της αγοράς. Κάποια κράτη-μέλη θα κάνουν δικές τους προτάσεις και δεν τα κατηγορώ γι' αυτό. Δεν είναι μόνο γι' αυτό το λόγο που χρειαζόμαστε ένα αποτέλεσμα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διεθνή συζήτηση και ευρωπαϊκή προσέγγιση. Κάτι που έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βραχυπρόθεσμα. Έχουμε το DST, τη φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών και τον ορισμό της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας και το CCTB. Αυτή είναι η προσέγγιση ευρωπαϊκή. Μέσω ευρωπαϊκής προσεγγίσεως μπορείς να επηρεάσει κατά πολύ τη διεθνή συζήτηση. Ο Αλένα Μασούρ δίκιο είχε με αυτό που είπε. Δηλαδή, δεν πρέπει να περιμένουμε για τη ΣΥΠΑ να κάνουμε μια πρόταση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε για μια διεθνή λύση, διότι υπάρχουν διαφορές. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή προσέγγιση και να τους πρόξουμε αυτούς, να προωθήσουμε τη διεθνή συζήτηση. Και είπα, ε, δρούν μονομερός το θέμα αυτό για η νομοθεσία για τις περικοπές και λοιπά δεν συζητήθηκε ε, με την Ευρώπη. Χρειάζεται ευρωπαϊκή προσέγγιση. Πρέπει να ηγηθούμε. Ελπίζω σαν πρώτο βήμα προσωρινό μέτρο η φορολόγηση ψηφιακών υπηρεσιών, το DST, να τροφοδοτήσει συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο. Κάποια σχόλια. Έκκληση απευθύνω. Να αυξηθεί το πεδίο εφαρμογή. Το ζητά το κοινό. Να δούμε την Amazon, την Netflix, τις μεγάλες εταιρείες που μεγαλώνουν με ραγδαίο ρυθμό. Πρέπει να φορολογηθούν. Στο Συμβούλιο συζητούν το περιορισμό του πεδίου εφαρμογή και η πώληση δεδομένων να εξαιρεθεί. Αυτό είναι παράλογο. Ε. Εξε... Η πώληση των δεδομένων να εξαιρεθεί θα δημιουργήσει τεράστιο κενό κάτι τέτοιο στο φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Αυτό είναι σαφέστατο, ηλίου φαϊνότερο. Αξιολόγηση συνεπειών. Άκουσα αυτά που υπόθηκαν. Μιλάμε για ισότιμους όρους και δίκαιη φορολόγηση. Τρία τέταρτα το κουβεντιάζουμε και πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες των προτάσεων. Και κινούμεθα στα σκοτεινά, πρέπει να το δούμε αυτό. Είναι χαρτογράφητα ύδατα αυτά στα οποία κινούμεθα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι και αξιολόγηση είναι ποιο να κάνουμε δεν είναι ακριβή τα αποτελέσματα, αλλά χρειάζεται και πολιτική ερμηνεία και προσέγγιση να καταλήξουμε σε συμφωνία. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Να πετύχουμε μια καλή συμφωνία, όπως το κάναμε και με το CCTB και με το CCCTB. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Προθεσμία και για τις δύο εκθέσεις, για τις τραπολογίες στις 16 του μηνός στις 5 το απόγευμα. Ε, στις 19 Νοεμβρίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και αναμένεται να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας ΕΚΟΝ στις 3 Δεκεμβρίου με στόχο ε, να πάει στην Ολομέλεια και να ψηφιστεί το Γενάρη του 19 με το καλό. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα μέχρι να έρθει η Επίτροπος. Ευχαριστώ.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 Dear colleagues, good Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Να καλωσορίσω την Επιτροπό Ανταγωνισμού, Μάργκερετ Βεστάγκερ, για τον δεύτερο και τελευταίο δομημένο διάλογο για το 2018. Είναι μια εξαιρετή ευκαιρία να μιλήσουμε για πολιτική ανταγωνισμού, εξαιρετική ευκαιρία να εκφράσουμε την υποστήριξή μας, κύριε Επίτροπε, διότι αποδειχθήκατε εξαιρετικά δραστήρια και σύγχρονη θα έλεγα στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στον περιβάλλον, στο, στην παγκόσμια αγορά. Η πολιτική σας, η πολιτική μας θα βοηθήσει τους πολίτες και τους καταναλωτές. Φυσικά υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, όπως η υπόθεση του Λουξεμβούρου. Χαιρόμαστε για τα όσα κάνατε. Υπήρχε μη διπλή φορολόγηση, όμως ε, τότε συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να τροποποιήσουμε την ομοθεσία μας. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αν έγινε αυτή η τροποποίηση όντως και θα δούμε πώς με την πολιτική αναγωνισμού μπορούμε να προχωρήσουμε στο νομοθετικό τομέα βεβαίω για να προλάβουμε τέτοιου είδου ε, περιπτώσεις στο μέλλον. Ήταν καλή προσπάθεια, ανεξαρτήτως αποτελέσματο. Ε, κατανοούμε και τις νομικές δυσκολίες βεβαίως. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα λόγω της κείμενης νομοθεσίας. Φυσικά όλα αλλάζουν, αλλά καλό είναι να βλέπει κανείς λίγο φως στην άκρη του τούνελ χάρη στις δικές σας προσπάθειες. Φαντάζομαι θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να υπενθυμίσω που βρισκόμαστε, τι κάνουμε για θέματα πολιτικής ανταγωνισμού αυτή τη στιγμή. Είμαστε κοντά στην ψήφιση του Ίσιαν Συν. Επίσης, δουλεύουμε επί της εκθέσεως Λούνας. διαβουλεύσει για την εφαρμογή του, των άρθρων 107 και 108 και θα συζητήσουμε το θέμα το απόγευμα. Θα αποφασίσουμε και για την διαδικασία και για πρώτη φορά Δουλεύουμε για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει τις πολιτικές ανταγωνισμού. Αυτό είναι πολύ καλό για μας. Ο κ. Λούνς Σιτής θα υποβάλει την, το σχέδιο γνωμοδότησης στις 22 Οκτωβρίου και βεβαίως έχουμε και την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Ο κύριος Ρέιμον είναι ο εισήγητης. Έχει υποβάλει σχέδιο έκθεσης θα τη συζητήσουμε 18 Οκτωβρίου. Οπότε, η παρουσίαση εδώ είναι απολύτως επίκαιρη γιατί όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε την υπόθεση του Λουξεμβούργου, την Google και παρόμοιες εταιρείε. Προσβλέπουμε λοιπόν σε μια επικοδομητική συζήτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε, Μαρκρέτε. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή. Χαίρομαι που ενδιαφέρεστε, αλλά και που παίρνετε και θέση όσον αφορά την αξία των εισόδημων κανόνων των ίδιων μέτρων και σταθμών. Πολλοί νομικοί, οικονομολόγοι λένε ότι είναι υπερβολικά πολύπλοκη νομοθεσία. Ξέρετε, το θέμα είναι η απλούστευση. Όταν είναι απλές οι αγορές, τότε οι καταναλωτές θα επιλέγουν ελεύθερα όπου θα αγοράζουν. Οι επιχειρήσει πρέπει να τηρήσουν τους νόμους και με αυτή την προϋπόθεση θα καινοτομήσουμε αλλιώ η καινοτομία θα πάει αλλού. Θέλουμε λοιπόν μια καλή αγορά η οποία θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη σε μια δική κοινωνία και Προσβλέπω στη συνεργασία μας και με τον Μισελ Ρεμόν για την επόμενη έκθεση για τις πολιτικές συναγωνισμού. Όταν έχουμε ανοιχτέ αγορές, τότε οι καταναλωτές εξασφαλίζουν τις καλύτερες τιμές, υπάρχει κίνητρο για καινοτομία, έχουν κίνητρα οι επιχειρήσεις δηλαδή να καινοτομήσουν. Φυσικά είμαστε υπέρ του ανταγωνισμού και λαμβάνουμε πρακτικά μέτρα. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο η λειτουργία των αγορών. Πολλέ φορέ οι καταναλωτέ ανησυχούν για προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να επιλύσει η αγορά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν από τι αγορέ να λύσουν τα πάντα. Και εκεί χρειάζεται να νομοθετήσουμε. Χρειαζόμαστε νομοθετικά μέτρα για να βοηθήσουμε την κοινωνία μα Κάτι το οποίο το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Και δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι και τα εθνικά κοινοβούλια που αναζητούν αυτόν τον στόχο. Ξεκίνησε, όπω ξέρετε, μια έρευνα για πέντε μεγάλους, ε, μεγάλες, μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων στη Γερμανία. Συνεργαζόμαστε. Η υποψία μας είναι ότι όχι μόνο συνεργάζονται σε θέματα ασφάλειας, ε, η υποψία μας είναι ότι προσπαθούν να αποφύγουν τον ανταγωνισμό σε θέματα τεχνολογικά που αφορούν τις εκπομπές κινητήρων, πετρελοκινητήρων και βενζινοκινητήρων. Εάν αποδειχθούν αυτές οι κατηγορίες, ε, τότε αυτό το οποίο θα έχει συμβεί ε, θα είναι ότι αυτές οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν απαγορεύσει ουσιαστικά ε, στους καταναλωτές να επιλέξουν καθαρότερα αυτοκίνητα. Ακριβώ επειδή αυτέ οι βιομηχανίες δεν χρησιμοποίησαν καθαρότερες τεχνολογίες που είναι ήδη διαθέσιμε. Ο ρόλος μας είναι να εξετάσουμε και να ερευνήσουμε προσεκτικά εάν η αυτοκινητοβιομηχανία, η αγορά αυτοκινήτου, εν τέλει λειτουργεί ελεύθερα υπέρ των καταναλωτών. Και εδώ χρειαζόμαστε καλή νομοθεσία για να μειώσουμε τις βλαβερές εκπομπές, εν γέννη, από τα οχήματα. Την περασμένη εβδομάδα, όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο υπερψήφισε νέου κανόνε για τι εκπομπέ οχημάτων. Η Κομισιόν εννοείται θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για να πετύχουμε του φιλόδοξου στόχου μα. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τι έρευνε περί κρατικών ενισχύσεων. Εδώ οι κείμενοι κανόνε απαγορεύουν στα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν αθέμητα πλεονεκτήματα στους λίγους. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και αθέμητες φοροαπαραγές, φορολογικά πλέον εκτίματα. Το 14, 15 δισεκατομμύρια πληρώθηκαν από 40 εταιρείε χάρη σε εμάς. Μια μεγάλη και κάποιες μικρότερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Όμως την φοροαποφυγή βάσει κανόνων κρατικών ενισχύσεων μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε ε, αν διαπιστωθεί η παράβαση. Γιατί ξέρουμε ότι κάποιες ε, επιχειρήσει κάποιες ε, αυτοκινητοβιομηχανίες μεταξύ άλλων απολάβουν αθέμητων πλεονεκτημάτων. Αλλά δείτε και σε άλλους τομείς, την McDonald's. Η McDonald's στο Λουξεμβούργο έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αθέμητα τη συμβασή αποφυγής διπλής φορολογίας με τις ΗΠΑ για να μεταφέρει κέρδη. Τα κέρδη όμω αυτά δεν φορολογήθηκαν τελικά ούτε στις ΗΠΑ ούτε στο Λουξεμβούργο. Τα συνδικάτα επέστησαν την προσοχή μας στη συγκεκριμένη κατάσταση. Και είναι πολύ καλό το ότι πολίτες, ε, ΜΚΟ και άλλοι ενδιαφέρθηκαν για το ζήτημα. Δημιουργήσαμε ενδελεχή ανάλυση που δεν επιβεβαίωσε όμως τις μέσα μας Δυστυχώ, Δυστυχώς ε, η συνθήκη επέτρεπε αυτήν την ειδική μεταχείριση. Ε, η McDonald's δεν ε, απείλευσε ειδικού μόνο για την εταιρεία και άλλε εταιρείε στην ίδια θέση. Οπότε τελικώ η McDonald's δεν παρεύει την νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίω ότι όλα καλά και άγια. Δεν είναι αποδεκτό ότι οι McDonald's ή οι επιχειρήσεις σε θέση μπορούν να εκμεταλλεύονται τις διαφορές στους φορολογικούς κανόνες μεταξύ ας πούμε, Χώρα ευρωπαϊκής χώρας και των ΗΠΑ για να μην πληρώνουν τελικά φόρο. Οπότε χαίρομαι που εν τέλει η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου θέσπισε νέα νομοθεσία για να διορθώσει την κατάσταση. Και αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο η McDonald's αλλά και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στην ίδια θέση ε, θα πληρώνει πλέον βάσει της νέας νομοθεσία. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που μας δείχνει γιατί πρέπει να συνδυάσουμε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων με άλλα επιπλέον μέτρα στον τομέα της φορολογίας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε λοιπόν εθνικά, ενωσιακά μέτρα και κανόνες για να εφαρμοστούν ίσα μέτρα και σταθμά για όλους. Έχει σημειωθεί ήδη σημαντική πρόοδος, χάρη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως απαιτούνται περισσότερα. Και βεβαίω πρέπει οι νέοι κανόνες όχι μόνο να υπερψηφίζονται, αλλά και να εφαρμόζονται από τις φορολογικές αρχές. Το προσωπικό τους, τα στελέχη, πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες και να τους εφαρμόζουν στην πράξη. Θα ήθελα σήμερα να σας διαβεβαιώσω ότι το έργο μας στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων θα συνεχιστεί. Προχωρούμε και με άλλε υποθέσεις. Υπάρχουν ε, κρατικέ ενισχύσεις με τη μορφή φοροαπαλλαγών ή άλλων πλέον εκτιμάτων. Διεργούμε επιπλέον έρευνες και αν υποπτευθούμε ότι αυτές οι ειδικέ μεταχειρήσει ε, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, θα παρεύουμε. Φυσικά, οι αγορές μπορούν να υπηρετήσουν τους πολίτες ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα στην ψηφιακή εποχή. Εδώ το θέμα είναι η Google και οι παράνομε συμπεριφορέ τη. Η Google εκμεταλλεύτηκε την. Ε, καταχράστηκε τι ε, δεσπόσε θέσει τη ε, σε πουλιστέ, τάμπλετ κλπ. Είναι η μηχανή που χρησιμοποιούν δισεκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα. Πιστεύουμε ότι ο στόχος τη Google ήταν να ενισχύσει τη θέση της στις επιγραμμικές αναζητήσεις. Αυτό που κάνουμε κάθε μέρα μέσω του τηλεφώνου μας ή του τάμπλετ. Οι κατασκευαστέ τηλεφώνων που ήθελαν να προσφέρουν το Play Store έπρεπε να προεγκαταστήσουν την, το Google και τον Chrome, τη μηχανή αναζήτησης. Και ήθελε μάλιστα η Google να το κάνει αυτό ε, χωρί επιτρέψει, απαγορεύοντα την εγκατάσταση άλλων προγραμμάτων. Επέβαλε λοιπόν τις δικές, δική τη μηχανή αναζήτηση σε συγκεκριμένε συσκευέ. Επίση, οι εταιρείε ε, που παράγουν τα τηλέφωνα και με Android πρέπει να ζητήσουν σχετικέ ε, άδειε από την Google. Η Google λοιπόν έκλεισε την αγορά. Η Google αποφάσισε ποιο λειτουργικό σύστημα, ποια μηχανή αναζήτησης ε, θα εγκατασταθεί στην οποιαδήποτε αγορά. Όμως εμείς θέλουμε μια ανοιχτή ε, αγορά. Θέλουμε να μην επιλέγει η Google αλλά οι καταναλωτέ να κάνουν ελεύθερη την επιλογή τους. Οπότε το πρόστιμο για την Google είναι πάνω από 4 δισεκατομμύρια και ζητήσαμε από την ε, Google να σταματήσει την παράνομη συμπεριφορά. Θέλουμε οι ανταγωνιστές της Google να έχουν ίσες ευκαιρίες να προσεγγίσουν τους καταναλωτές με συσκευέ βάσει του λειτουργικού Android και περισσότερες επιλογές σημαίνει περισσότερη καινοτομία. Έτσι, οι εταιρείε ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών θα μπορούν να αξιοποιούν τι μηχανέ τη Google και του Android, αλλά θα μπορούν να αναπτύξουν και τι δικέ του εφαρμογέ ε, πάνω στα μέσα αυτά. Η περί ανταγωνισμού νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν να είναι και αυτή έτοιμη για την νέα ψηφιακή εποχή. Πολλά πράγματα έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί, όμως βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή αυτής της ψηφιακής επανάστασης. Τον Μάρτιο όρισε τρεις ειδικού συμβούλους για να εξετάσουν την κατάσταση στην αγορά. Ο ένας ε, ξέρει τα οικονομικά, ο άλλος ξέρει τον ανταγωνισμό και ο τα τεχνολογικά. Θέλουμε να εξακριβώσουμε κατά πόσον οι κανόνες μας ανταποκρίνονται στι ανάγκε της νέας ψηφιακή αγορά. Οι τρεις ε, σύμβουλοι και εγώ θα φιλοξενήσουμε μία διάσκεψη τον Ιανουάριο. Θέλουμε φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε όλη αυτή την προσπάθεια από την πλευρά μα, Η κατάσταση της Ένωσης χαρακτηρίζεται από ταχύτερες εξελίξει θέλουμε να δούμε πού και πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία, που υπάρχουν προβλήματα και πώς θα τα επιλύσουμε. Με ίδια ορμητικότητα, με την ίδια όρεξη προτείνουμε ω Κομισιόν κανόνες εκεί που λείπουν για να προστατεύσουμε μεταξύ άλλων το περιβάλλον. Ε, οι χώροι εργασία να γίνουν ασφαλείς χώροι εργασία. Είναι συνδυασμό ε, ανταγωνισμού, και προσπάθεια εφαρμογή τη νομοθεσία για μια καλύτερη Ευρώπη. Προσβλέπω σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι ξέρω πώ λειτουργεί το όλο πράγμα και πραγματικά πρέπει να προχωρήσουμε μαζί προς τα εμπρό σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ε, εντάξει, νομίζω ότι θα έχουμε καλές ερωτήσεις μετά την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ που υπογραμμίσατε πολύ καλά το θέμα της υποθέσεως Μακδόναλτ στο Λουξεμβούργο. Προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση της νομοθετικής αυτής επανεξέτασης και ελπίζω ότι με το κείμενο CCTB που θα εθετηθεί από το Συμβούλιο ε, θα βοηθήσουμε να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό δείχνει τα ωφέλη ενός πλαισίου νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποφεύγει αυτή τη φορολογική αποφυγή, τη διπλή μη φορολόγηση Σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε με τον πρώτο μιλητή. Ο Ανδρέας Σφάμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Νομίζω ότι ήταν πολύ συναρπαστική η εισαγωγή. Κάνατε μια ηθατή επισκόπηση όλων των θεμάτων και σε σχέση με αυτό που μόλις είπε ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη, η τελική ψηφοφορία ε, από το Κοινοβούλιο ε, επίκειται και δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, οπότε μπορώ να έρθω σε άλλα θέματα που μας περιμένουν. Ε, να επανέλθω λίγο στις κρατικές ενισχύσεις ε, ως εργαλείο ελέγχου της φορολογικής πολιτικής των κρατών μελών. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό το εργαλείο και πολύ συχνά δέχεται επικρίσεις από πολλούς συναδέλφους, όχι μόνο στις εθνικές βουλές, για τα αποτελέσματα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, αποδείχθηκε αποτελεσματικό εργαλείο που δείχνει ότι στην Ευρώπη εργαζόμαστε υπέρ ε, ίσων κανόνων και θεμητού ανταγωνισμού προς όφελος όλων των πολιτών. Και χρειαζόταν θάρρος πραγματικά για να επιβληθεί αυτό εις βάρος κάποιων κρατών μελών που είχαν ε, άσχημη συμπεριφορά όχι μόνο προς τους γείτονές τους αλλά και έδιναν και φορολογικά κίνητρα ή ε, κίνητρα φοροαπαλλαγών ε, σε κάποιες εταιρείες οι οποίες τα εκμεταλλεύτηκαν και ε, κατεστάθηκαν και χάθηκαν και φορολογικά έσοδα προς όφελες των πολιτών. Είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε τους συναδέλφους στα κράτη-μέλη και μπράβο σας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για κάποιες άλλες περιπτώσεις που αναφέρατε. Διάβαζα στο Sky News δεν ξέρω πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το νέο εχθές, ότι προσπαθεί η Google να αποφύγει, να παρακάμψει οι κανόνες στην Ευρώπη ε, με διάφορες άλλες ε, μεθόδους. Ισχύει αυτό. Και τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι δράση θα αναλάβει κατά της εταιρείας. Και επόμενη ερώτηση για το Brexit γιατί στον έλεγχο των συγχωνεύσεων έχουμε μπροστά μας συγχώνευση Disney ε, με τη Fox. Ε, τι θα γίνει αν έχουμε σκληρό Brexit, γιατί διάφορα ζητήματα θα συνδεθούν με το ζήτημα αυτό. Αν θα παραμείνει η αγορά, η συγχώνευση θα ε, να βαγίσει. Και χαίρομαι που ε, Προτείνετε να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στα όσα θα συζητήσετε για τον ανταγωνισμό στην ψηφιακή οικονομία και εποχή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για το έργο που κάνατε. Προσβλέπω λοιπόν στην ψηφοφορία και ήδη συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να προετοιμαστούμε για το N+, να εφαρμοστεί στη διεθνή νομοθεσία ούτως ώστε οι πολίτες να ωφεληθούν ε, πλήρως από το έργο που έχει γίνει για να μπορούν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού να τους προσέξουν σε εθνικές αγορές. Νομίζω ότι αυτό το κοινοβούλιο έκανε υπέροχη δουλειά και βέβαια με εσά ως εισηγητή επιταχύνεται νομοθετική διαδικασία. Και αυτό ήταν εντυπωσιακό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των διαφημιστικών εταιριών και αυτό μας έχει ε, το έχουμε προσέξει ε, ε, ψευδείς συγκρίσεις ιστοσελίδες που κάνουν ψευδείς συγκρίσεις και θέλουμε να δούμε πώς εξελίσσεται η αγορά είναι δούριος ύπος για να γίνουν κάποιες αλλαγές το εξετάζουμε για έλεγχο συγχωνεύσεων και το Brexit σε κάποιο βαθμό Έχουμε σχεδιασμό για έκτακτες περιστάσεις. Από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει κενό μεταξύ της ημερομηνία του Brexit και της ε, έναρξης της σωστής κάλυψης. Ε, νομίζω ότι θα υπάρξει πολύ καλή συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν πάρα πολύ καλό πνεύμα για τον ανταγωνισμό και πολύ καλούς αρμόδιους φορείς και δημιουργούμε σχέσεις για να συνεχιστεί η σωστή προσέγγιση όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε και για τη δέσμευση που αναλάβατε για να κάνετε την πολιτική ανταγωνισμού μια πολιτική που θα προστατεύει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Λυπούμε που δεν μπορέσετε να καταλήξετε σε πιο επιχειρησιακά ε, συμπεράσματα. Καταλαβαίνουμε όμως αυτά που μας είπατε. Και αν εντοπίζετε τα κενά στην νομοθεσία, αυτό είναι καλό. Αυτό δείχνει τα όρια της πολιτικής ανταγωνισμού όσον αφορά την κάλυψη των κενών στη φορολόγηση. Αυτή η περίπτωση ολοκληρώνει τις έρευνες για τις αποφάσεις για τα φορολογικά, για τα tax rulings ή έχετε κάποιο απόθεμα θεμάτων προς εξέταση. Το tax ruling σας και tax planning practice αποτελεί αντικείμενο εξεργασίας ακόμα. Άλλη μια ερώτηση. Για την κατάσταση που επικρατεί στη Μαδέιρα. Εκεί προβληματίζονται οι Πορτογάλοι φίλοι μας για τα φορολογικά προνόμια της νήσου. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, τι γίνεται. Υπάρχουν κενά. Θα ξέρετε για αυτό το θέμα. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Θα ήταν καλό. Τρίτον, την οριζόντια προσέγγιση που προτείνεται για τον ανταγωνισμό στον ψηφιακό τομέα. Πώς διαθρώνεται αυτή η προσέγγιση και ο προβληματισμός με μια άλλη πτυχή που σας ανησυχεί πολύ και σας προβληματίζει. Αυτή σχετίζεται με, τον ιδιωτικό, με την ιδιωτικότητα των δεδομένων, με προσωπικά δεδομένα, πώς προστατεύονται αυτά και ο ψηφιακό κόσμος πώς μπορεί να ταιριάξει με την ιδιωτικότητα και τα ατομικά στοιχεία. Αυτά πώς θα συμπεριλαμβάνετε στο γενικότερο προβληματισμό σας για το μέλλον του ανταγωνισμού στον ψηφιακό τομέα. Απάντηση. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τη μεγάλη υποστήριξη που έχετε δώσει όσον αφορά το έργο μας όταν εξετάζουμε κατά πόσο καταβάλλεται παράνομη κρατική ενίσχυση. Ζητάμε από όλα τα κράτη-μέλη να μας πούν πώς χρησιμοποιούν τις αποφάσεις τα τα tax rulings. Έχουμε πάρει στοιχεία από τα κράτη-μέλη, παίρνουμε ένα δείγμα από τα στοιχεία των κρατών μελών. Τι είναι οι εταιρείε πολυεθνικές, μη πολυεθνικές κλπ. για να έχουμε πλήρη εικόνα. Ποια είναι τα καλά νέα, ότι τεράστια πλειοψηφία των κρατών μελών Εάν ε, εφαρμόζουν τα tax rulings, το κάνουν καλά. Υπάρχει σωστή τεκμηρίωση για τις αποφάσεις, τιμές που είναι πολύ κοντά στις τιμές της αγοράς, οπότε είναι καλή δουλειά που κάνουν. Πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εξέταση του θέματος και ίσως να δώσουμε και κάποιες ιδέες γραπτός σχετικά με τα μαθήματα που έχουμε ε, αντλήσει από όλα αυτά. Τούτου λεχθέντος Έχουμε ερωτηματολόγια που έχουμε αποστείλει, γιατί ίσως χρειάζονται και άλλες προσφυγές. Και αυτό είναι μονίμως ένα πρόβλημα. Και έχει, έχουμε την Task Force για τα φορολογικά, η οποία έχει μετατραπεί σε μία μόνιμη μονάδα στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Comp, για να συνεχιστεί το έργο. Έχουμε κάνει πρόοδο βέβαια, όμως είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι θα συνεχίσουμε να ενδιαφερόμαστε για το κατά πόσο υπάρχει συνεχής πρόοδο στον τομέα ή όχι. Το θέμα της Μαδέρα. Συνεχίζονται οι, ε, οι διαβουλεύσεις και η εξέταση του θέματος. Αν θέλουμε ειδική κάλυψη για τη Μαδέρα και να δούμε αν αυτές οι, αυτές οι διατάξεις περί Μαδέιρα αν τις εκμεταλλεύονται. Δηλαδή ισχύουν κάποια πράγματα για τις ιδιαίτερες περιστάσεις του νησιού, αλλά πρέπει να αναγνωρίζονται. Αν έχεις ένα ειδικό μηχανισμό που δεν διατίθεται στην υπηρετική Ευρώπη για να δημιουργήσει θέσει εργασία ή για να προσελκύσει επιχειρήσεις, το χρειάζεσαι γι' αυτό και όχι να δημιουργήσει εταιρείε εικονικέ γραμματοκιβωτίου, διότι αυτό δεν δημιουργεί θέσει απασχόλησης, εικονικές εταιρείε. Εξετάζουμε το θέμα, θα δούμε αν οι υπόνοιέ μα τελικά αποδειχθούν ότι ευσταθούν, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό όταν θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για τα δεδομένα τώρα. Όταν ελέγχουμε συγχωνεύσεις, εξετάζουμε συνήθως τι είδου στοιχεία συγχωνεύονται όταν συγχωνεύονται εταιρείε ιδιωτική φύσεω που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χρήσουν ιδιαίτερη προσοχή, παράγουν δεδομένα που θα χαθούν και πρέπει την επομένη να επανεξεταστούν. Αυτά τα δεδομένα δεν έχουν αξία. Δεδομένα που προέρχονται από συμπεριφορά πελατών που δεν είναι προσωπική φύσεω αλλά πολύτιμα στοιχεία όσον αφορά την καινοτομία, πηγέ για καινοτομία. Και μετά είναι φραγμός. Είναι πολύ δύσκολες, είναι δύσκολο για άλλε επιχειρήσεις μετά τη συγχώνευση να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Δεν είχαμε περίπτωση όπου να έχουμε πρόβλημα με τα δεδομένα και να μας ενοχλεί αυτό για τη συγχώνευση. Συνήθως στην ανάλυση τα συμπεριλαμβάνουμε τα στοιχεία και εμβαθύνουμε στην ανάλυση ε, της ψηφιοποίησης. Δεν θυμάμαι συγχώνευση που να μην έχει μια ψηφιακή πτυχή και πτυχή ε, δεδομένων. Το είδαμε στη συγχωνεύση στον αγροχημικό τομέα. Η ψηφιακή γεωργία προωθείται στην υγεία. Παντού το βλέπουμε. Διότι αυξάνονται οι πωλήσει που ακολουθούν επιτρέπεται να γίνουν βελτιώσεις και σου επιτρέπει να παραμείνει στην αγορά με διαφοροποίηση. Και συνεχώ θα το βρίσκουμε μπροστά μα αυτό. Γιατί όσον αφορά τα δεδομένα, αυτά τα χρόνια που περνάνε, ε, συνεχώς μεταλλάσσεται η προσέγγιση. Ευχαριστώ, ο Ραμόν Τρεμόσα. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Αγαπητοί Επίτροπε, καλώ ορίσατε και πάλι στο Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ για όλη τη καλή δουλειά που κάνετε και υπερασπίζεστε του Ευρωπαίου καταναλωτέ, το θεμητό ανταγωνισμό και το εγχείρημα τη ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Και θα χαρώ να συμμετέχω κι εγώ στο εργαστήριο, στη διάσκεψη που είπατε για τον Ιανουάριο, για την Google. Πριν από 8 χρόνια ξεκίνησε επί Επιτρόπου Αλμούνια αυτή η προσπάθεια. Σήμερα πού βρισκόμαστε και πότε ε, θα αναμένατε την τελική απόφαση πριν φύγετε, πριν λήξει η σας. Την τελευταία φορά που ήρθατε είπατε ότι είδατε κάποιες βελτιώσεις της μηχανής αναζήτησης. Μπορείτε να, το επιβεβαιώσετε. Δεύτερη ερώτηση για την Αλιτάλια. Μπορείτε να μας δώσετε μια ενημέρωση τι έχει μεσολαβήσει εκεί. Η νέα Ιταλική κυβέρνηση απάντησε για τις προθέσεις της ε, αναδιάρθρωσης της εταιρεία. Έχει πάρει 900 εκατομμύρια δάνειο γέφυρα. Έχει πληρώσει Τόκου. Μετά, συγχώνευση Siemens με την Alstom. Έχει τεράστιες επιπτώσεις για το σιδηρόδρομο στην Ευρώπη αυτό. Ποιες είναι οι συνεισφορές ε, που έχετε λάβει από μικρότερους φορείς της αγοράς. Η Alstom και η Siemens μαζί θα καλύπτουν το 80% των σιδηροδρόμων στα κράτη-μέλη και το τροχιοελικό μηχανές και συστήματα σημάτων. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό συνάδει με την ε, ελεύθερη αγορά. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη σας ερώτηση. Αυτή η ιστορία με την Google ε, πάει μια οχταετία τώρα. Θα πρέπει να το δούμε και να καταλάβουμε γιατί πρέπει να μπορούμε να λύνουμε μια υπόθεση με διάφορους τρόπους μπορούμε, έχουμε διάφορες διαδικασίες. Ε, με, η απαγόρευση και το πρόστιμο είναι το τελευταίο. Μπορεί να γίνει και με συνεννόηση και με ε, επίλυση διαφοράς. Αν μπορούσε να είχε λύσει την υπόθεση η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν καλύτερα φυσικά, γιατί θα είχε λυθεί νωρίτερα και κάποιες από τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την παράνομη συμπεριφορά της Google θα είχαν ανθίσει γιατί θα λειτουργούσε καλύτερα η αγορά. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Εξού και επιλέγει άλλος δρόμος. πού βρισκόμαστε σήμερα. Διαπιστώνουμε ακόμα κάποιες αλλαγές στους ανταγωνιστές του Google Shopping, ε, αλλά προσέχουμε πάρα πολύ να μην παρασυρθούμε από τους αριθμούς για να καταλήξουμε σε λάθος συμπεράσματα. Το θέμα δεν είναι πόσες μηχανές υπάρχουν, ε, αλλά πώς λειτουργεί η αγορά και πώς ε, τοποθετούνται αυτές οι μηχανές αναζήτησης και οι ανταγωνιστές. Όλοι έχετε και έχουμε ε, καταλάβει ότι δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε οριστική θέση, άρα είναι ανοιχτή η έκβαση. Για το δεύτερο ερώτημα, σχετικά με την Αλιτάλια και τα σχέδια της Ιταλικής κυβέρνησης. Δεν έχω καμία ενημέρωση σχετικά. Η υπόθεση τρέχει ακόμα και θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το επίπεδο των τόκων που θα πρέπει να καταβληθούν. Στο παρελθόν είδαμε σε περίπτωση κρατικών ενισχύσεων ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το ζήτημα αυτών των τόκων, το ακριβές μέγεθος. Γιατί αν μπορεί μια κυβέρνηση να επενδύσει σε μια εταιρεία, ε, έχει σημασία το, το επιτόκιο γιατί αλλιώς ε, μπορεί να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση. Για ε, την Alstom ε, Siemens πολύ γρήγορα μας τράβηξε την προσοχή. Ακόμα ήταν άτυπη αυτή η διαδικασία. Έχουν αρχίσει διάφοροι να έρχονται και να μας κάνουν κρούση ότι κοιτάξτε θα γίνει κολοσσός η εταιρεία αυτή στην Ευρώπη. Εμείς τι αναλύουμε ποιο ρόλο παίζουν στην ευρωπαϊκή αγορά άλλες παγκόσμιες μεγάλες επιχειρήσεις. Θα αυξηθούν οι τιμές, θα μειωθεί η επιλογή για το τροχαίο υλικό και τα σήματα στην Ευρώπη λόγω της συγχώνευσης. Ε, πώς θα επηρεάσει αυτό τις άλλες εταιρείες για τις εμπορευματικές ε, και επιβατικές μεταφορές. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ανάλυση, αλλά ελπίζουμε Όποιο ανησυχεί να έρθει να μα το πει. Δεν είναι ακόμα πολύ αργά. Αν κάποιο ανησυχεί για τη συγχώνευση αυτή και την αγορά των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη, που είναι ιδιαίτερη αγορά και παγκοσμίω. Γιατί το δίκτυο είναι πάρα πολύ παλιό. Αλλά ε, ελάτε, αν έχετε κάποιες ανησυχίες, με χαρά να τις ακούσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, ασχητής. Ε, Κύριε Επιτροπέ, καλώς ήλθατε. Χαίρομαι να συνεργαζόμαστε, γιατί έχετε μια πολύ σαφή εικόνα περί του πώς πρέπει να είναι η πολιτική ανταγωνισμού. Να λειτουργεί η αγορά για τους καταναλωτές και για τις ανταγωνιζόμενες εταιρείες. Περί αυτού πρόκειται. Και ξέρω ότι αυτό επιδιώκεται. Οι άλλοι στόχοι δεν είναι ανταγωνισμό. Άλλο η μεταβολή του κλίματος και ούτω καθεξής. Άλλο η κοινωνική δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ναι στους νόμους που πρέπει να διέπουν την πολιτική ανταγωνισμού. Αυτό με βρίσκει βεβαίως σύμφωνο. Τώρα, όταν μιλούμε όμως για ψηφιακή αγορά, βρισκόμαστε και πάλι αντιμέτωποι το εξή πρόβλημα. Αν η αντιμετώπιση περιοριστεί στην νομοθέτηση, θα τρέχουμε πάντα πίσω από τις εξελίξεις. Γιατί η θέσπιση, η υπερψήφιση, η ενημέρωση της νομοθεσίας κρατάει 10 χρόνια και η αγορά θα έχει πάει αλλού. Όταν ξεκίνησε, η Ευρώπη ξεκίνησε την πολιτική ανταγωνισμού, το θέμα δεν ήταν μόνο η προστασία των καταναλωτών και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ήταν ο περιορισμός της υπερβολικής επιρροής κάποιων επιχειρήσεων. Το πεδίο αυτό το αντικείμενο αυτό διευρύνεται ακόμη περισσότερο στις μέρες μας, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ψηφιακές επιχειρήσεις όπως η Google, η Microsoft, το Facebook και άλλε. Τι γίνεται όταν αυτοί χρησιμοποιούν τα στοιχεία μου, τα προσωπικά μου δεδομένα. Ε, φοβούμαι ότι με χρησιμοποιούν ως χρήστη και όχι ως καταναλωτή. Το πράγμα ξεφεύγει από την πολιτική για τους καταναλωτούς και καταναλωτές, η προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική. Ξεφεύγουμε λοιπόν από την πολιτική ανταγωνισμού και εννοείται ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εμεί ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσουμε το θέμα ευρύτερα. Για παράδειγμα, έχουμε έναν υποψήφιο από το ΕΛΚ, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει πρόεδρος της επόμενης Κομισιόν και ο οποίος είπε ότι το Facebook πρέπει να το μεταχειριστούμε διαφορετικά και έχω πρόβλημα εκεί. Στην έκθεση περί ανταγωνισμού, όταν μιλάμε για μια διευρυμένη αντιμετώπιση των θεμάτων ανταγωνισμού, ενόψη του μέλλοντος, για το πώ θα συνεργαστούμε, ε, εσείς ως φιλελεύθεροι, πώς το βλέπετε. I think to... Έχουμε εδώ δύο διαφορετικά πράγματα. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι περιχαρακωμένη, περιδιαγεγραμμένη με διάφορους τρόπους. Και αυτό είναι καλό. Δηλαδή έχουμε δημοκρατία στην Ευρώπη, στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνουμε αποφάσεις για το περιβάλλον, για τις συνθήκες εργασίας, για την παιδική εργασία και ούτω καθεξής. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν λέμε κατά τα άλλα, οκ, βγείτε έξω στον ανταγωνισμό με βάση όμως κανόνες. Γιατί κανείς νομίζω δεν θα αποδεχόταν μια ελεύθερη αγορά χωρίς κανόνες. Δεν θα έχει κανένα νόημα αυτό. Ακόμη περισσότερο σήμερα που τέτοιες εξελίξεις, κάθε άλλο παρά σε ελεύθερη αγορά, θα οδηγούσαν θα είμαι μια αγορά μονοπωλίων. Αυτό είναι μια πτυχή, μια πλευρά. Και επαναλαμβάνω ότι έχουμε και ανταγωνισμό και κανόνες. Και ανταγωνισμό και νομοθεσία. Γιατί αυτό απαιτούν οι δημοκρατίες μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις στην ελεύθερη αγορά. Τώρα, Όλα αυτά εξελίσσονται. Μιλούμε πολύ για παράδειγμα για δεδομένα. Γιατί ξέρουμε ότι, ε, ξέρουμε ότι τα δεδομένα είναι μια πρώτη για την καινοτομία, ξέρουμε ότι είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, ξέρουμε ότι είναι ένα νόμισμα, ένα μέσο ανταλλακτικό αν θέλετε και η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να ακολουθήσει και αυτή, δηλαδή τα νέα αυτά ζητήματα. Θέλουμε καινοτομία βεβαίως, ο ανταγωνισμός εδώ είναι εργαλείο ε, και εμείς ακολουθούμε βήμα προς βήμα. Ας πούμε για τα αυτοκίνητα. Το καρτέλ της αυτοκινητοβιομηχανίας ε, είναι ένα καρτέλ καθορισμών ε, όχι τιμών πλέον. δεν είναι ούτε διαίρεση των αγορών. Εσύ θα πουλάς το βορρά και εγώ στο νότο. Όχι, είναι ένα καρτέλ το οποίο αποφάσισε να μην αξιοποιήσει την βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία για τις εκπομπές. Αυτό είναι καινοφανέ. Ε, αυτό είναι ένα καινοφανέ καρτέλ. Δεν είναι όπω παλιά που κάποιοι συμφωνούσαν ε, σε τι τιμέ τα πουλάνε. Θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμα και το πλαίσιο που περίγραψα αλλάζει και αυτό. Γιατί αλλάζουν οι πρακτικέ. Οπότε να ξέρετε ότι και εμεί δεν ε, καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Τροποποιούμε την νομοθεσία, την κείμενη νομοθεσία αυτήν που εφαρμόζουμε σήμερα και την τροποποιούμε γιατί αλλάζει η αγορά γύρω μας. Και έχουμε παραδείγματα επιτυχίας. Σε πολλές περιπτώσεις ε, αξιοποιήσαμε την κείμενη νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τετριμένα όπως ε, τα καφοπίστρα που είναι ξυλουργοί ε, και φτάνουν όλα αυτά μέχρι το, το Google Chrome και την ψηφιακή τεχνολογία. Βλέπετε λοιπόν ότι η κείμενη νομοθεσία είναι αρκετά ευέλικτη. Φυσικά πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται για να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες προκλήσεις. Για το τελευταίο που είπατε, πώς θα κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα αυτές τις τεράστιες εταιρείε, το πώς δημιουργούν αξία και να δούμε αν υπάρχει χώρος για άλλους, αν αφήνουν χώρο για άλλου. Μια λοιπόν συζήτηση που πρέπει να κάνουμε είναι εξή. Ξέρουμε πλέον ότι είμαστε κύριοι των προσωπικών μας δεδομένων. Τι κάνω όμω με αυτά τα δεδομένα. Μπορώ να τα δώσω σε κάποιον. Πώς. Θέλω να τα δώσω. Να τον διευκολύνω γιατί αν τα δώσουμε όλα όλοι μας τότε τα στοιχεία αυτή, αυτά θα είναι δεδομένα ε, στη διάθεση και επιχειρήσεων που καινοτομούν, αλλά υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις. Πρέπει να σταθμίσουμε αυτές τις επιπτώσεις. Τι γίνεται με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, στην... Πρέπει να έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Πρέπει κάποιες ε, επιχειρήσεις να διαιρεθούν, πρέπει να διευκολυνθούν, πώς θα ανταλλάσσουν δεδομένα με τρόπο δίκαιο στην αγορά, ώστε να υπάρχει και χώρος και πρόσβαση για τις άλλες ψήφικες εταιρείε. Ε, δεν έχω καταλήξει φυσικά συμπεράσματα ακόμη, γιατί ε, νομίζω θα, θα έπρεπε να ανησυχείτε αν είχα καταλήξει συμπεράσματα. Ε, χρειαζόμαστε πολλούς ειδικού οι οποίοι θα διερευνήσουν την κατάσταση, θα μελετήσουν την αγορά, θα χρειαστεί χρόνος, θα χρειαστεί να συζητήσουμε μαζί και βεβαίω η πολιτική και η νομοθεσία περί ανταγωνισμού είναι μια καλή αφορμή. Κύριος Παπαδημούλη. Ε, σας καλωσορίζω κυρία Επίτροπε. Ε, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας. Προτιμώ να μιλήσω ελληνικά. Ε, όπως είδατε ήδη για μια ακόμη φορά, στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει μια πολύ ευρεία και οριζόντια πολιτικά πλειοψηφία που στηρίζει τη δουλειά σας ως Επιτρόπου Ανταγωνισμού. Και ο λόγος είναι γιατί ε, σχεδόν όλοι εδώ μέσα συμφωνούμε με τη βασική ιδέα που μας παρουσιάσατε. Ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από τις αγορές να λύσουν τα πάντα. Χρειάζεται να νομοθετούμε. Να αξιοποιούμε την υπάρχουσα νομοθεσία ή και όπου έχουμε καινούριε προκλήσεις να βελτιώνουμε την νομοθεσία δεν είμαι βέβαιος αν έχετε ως αρμόδια επίτροπος για τον ανταγωνισμό την ίδια υποστήριξη και από τα κράτη-μέλη ή από αρκετά κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, όπως η υποστήριξη που έχετε από το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τρία πράγματα. Το πρώτο, επειδή όντω είναι πολύ σημαντικό και θα έλεγα επικίνδυνο να υπάρχει ένα καρτέλ αυτοκινητοβιομηχανιών που δεν κανονίζει μόνο τις τιμές αλλά ορθώνει και εμπόδια στο να αξιοποιείται τεχνολογία που εξασφαλίζει μικρότερους ρήπους, η οποία ήδη υπάρχει και επειδή μόλις την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωκοινοβούλιο εψήφισε με μια καθαρή, μεγάλη πλειοψηφία μια έκθεση που ζητά μια ταχύτερη, πιο φιλόδοξη μείωση των ρήπων, θα ήθελα να μας πείτε πότε εκτιμάτε ότι θα υπάρχουν κάποια αποτελέσματα της έρευνας που κάνετε, ε, γιατί όπως μας είπατε έχετε υποψίες ότι εκεί πέρα γίνεται κάτι που δεν είναι καθόλου καλό από αυτό το καρτέλ. Η δεύτερη μου ερώτηση. Είπατε ότι για τα tax rulings ε, η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών κάνει καλή δουλειά. Τεκμηριώνει με παραδείγματα ότι τα αξιοποιεί σωστά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την άλλη πλευρά του φεγγαριού. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχετε την αίσθηση ότι δεν κάνουν καλή αξιοποίηση των tax rulings, που δεν σας έδωσαν επαρκή στοιχεία, που νομίζετε ότι πρέπει να υπάρχει κάποια έρευνα ή τομείς ή παραδείγματα όπου τα tax rulings χρησιμοποιούνται όπως στην περίπτωση της McDonald's που μας είπατε ότι αποδείχθηκε ότι αυτό που γινόταν ήταν νόμιμο σε πολλά εισαγωγικά αλλά δεν ήταν καθόλου δίκαιο και καθόλου ηθικό και έστω και με καθυστέρηση η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου το άλλαξε. Και η τρίτη μου ερώτηση. Ε, επειδή διαβάζω και διάφορα δημοσιεύματα, είναι λίγο πιο προσωπική αυτή. Επειδή διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εσά και στα μελλοντικά σας σχέδια και τη δουλειά σας στην Κομισιόν. Θα σας ενδιέφερε, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της θητείας αυτής, να συνεχίσετε ως Επίτροπος ή ενδεχομένως και με έναν υψηλότερο ρόλο για τα θέματα που μας παρουσιάζετε. Είναι δύσκολο να πούμε πότε θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα στο καρτέλ των αυτοκινήτων, ε, στην ε, διερεύνηση. Αλλά ξέρουμε ε, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Κάθε στο αυτοκίνητό σου βάζεις το κλειδί και ε, καρτέλ είναι ακόμα και όταν βάζεις μπρος τη μηχανή, όταν ανάβεις τα φώτα, τα καθίσματα, ε, ε, πολλά στοιχεία του κινητή. Ξέρουμε πολύ καλά την αυτοκινητοβιομηχανία και πού ήταν τα καρτέλα, αλλά υπάρχει και εκεί η άλλη όψη του νομίσματος, διότι θέλουμε να συνεργάζεται η αυτοκινητοβιομηχανία για τα μέτρα ασφαλείας ε, ή ακόμα για να κάνουν το άλμα προς τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη χρήση των σόρευτων και την ανακύκλωση και τα λοιπά και πώς κατασκευάζονται οι μπαταρίες. Για να γίνει αυτό θέλουμε να προάγουμε τη συνεργασία μεταξύ κατασκευαστών αυτοκινήτων και άλλων επιχειρήσεων σε αυτή την αλυσίδα παραγωγής αξίας. Προσπαθούμε να είμαστε λοιπόν ε, ανοιχτή στην προσέγγιση μας. Δεν βλέπουμε παντού καρτέλ, αλλά μόνο εκεί που είναι επιζήμιο για μας ως καταναλωτές. Και όπως σας είπα για τις εκπομπές, αυτό είναι υπέρ των καταναλωτών και μάλιστα στην κυριολεξία. Το είπα και στην εισαγωγή. Χαίρομαι με την προσέγγιση του Κοινοβουλίου. Οι συνάδελφοι που ασχολούνται ε, ε, με αυτά τα θέματα ε, ρύθμισης για τους ρήπους και για το σχετικό σκάνδαλο είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Για τα κράτη-μέλη σχετικά με τα tax rulings και πού έχουμε κάποια ερωτηματικά. Κάνουμε ερωτήσεις στα κράτη-μέλη και εξακολουθούμε. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμίε υποθέσεις ακόμα. Έχουμε το θέμα του IKEA αλλά και κοιτάμε και τα διάφορα συστήματα που δεν είναι tax rulings, ε, αλλά που έχουν στηθεί κάποια συστήματα για ορισμένους λίγους και όχι για τους πολλούς ή για όλους. Το CFC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, ναι, ναι, Το Kentucky Fried Chicken. Εμείς ασχολούμαστε με τις ειδικέ περιπτώσεις, ενώ το Συμβούλιο περνάει νομοθεσία για να αλλάξει παγκοσμίω, ε, πανευρωπαϊκά συγγνώμη, ε, ελπίζω και ε, το προσεχώς το CCCTB, η κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση επιχειρήσεων, αλλά αλλάζουν και τα κράτη-μέλη τα ίδια. Ας πούμε η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου πέρασε καινούργια νομοθεσία, αλλά και στις κάτω άλλαξαν. Και στην Ιρλανδία αλλάζουν, στη Μάλτα, στην Κύπρο, δεν απατώμε και στην Κύπρο, αλλάζουν την νομοθεσία τους, έτσι ώστε ε, η εθνική νομοθεσία να ε, προσφέρεται καλύτερα και για να συνάδει με την ευρωπαϊκή. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Διότι έτσι βήμα-βήμα φτάνουμε πιο κοντά σε μια κατάσταση όπου δεν θα πληρώνουν τους φόρους οι περισσότερες εταιρείες, αλλά όλες οι εταιρείες. Και έρχομαι τώρα στο τελευταίο σας ερώτημα. Ε, το έχω ξαναπεί. Κάποιοι το ακούν, κάποιοι δεν θέλουν να τα ακούσουν. Ε, θέλω να ε, έχω άλλη μια θητεία ως επίτροπος και ή δυνατόν επίτροπος ανταγωνισμού. Ε, εγώ προσπαθώ να είμαι υπείων τόνων, αλλά θα έχετε διαπιστώσει ότι μου αρέσει η δουλειά μου και βρισκόμαστε στη μέση μιας προσπάθειας ε, έχουμε τους συμβόλους στις δικές σας ε, συζητήσεις, διασκέψεις, γίνονται καινούργια πράγματα. Ε, είμαστε στη μέση μιας διαδικασίας και θα ήταν τιμή όσο και προνόμιο για μένα να έχω την ευκαιρία να εξακολουθήσω να υπηρετώ τους Ευρωπαίους από το μετερίζει αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ε, θα μίλησω και εγώ στα ελληνικά. Ε, καταρχήν να συγχαρώ την Επίτροπο, γιατί θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε ένα δύσκολο περιβάλλον, ε, έχοντας μπροστά της να διαχειριστεί τεράστιες εταιρείε με, πολύ μεγάλες δυνατότητες. Θα ήθελα όμως να σας πάω λίγο, όχι τόσο στο μέλλον, που μπορεί να είναι ψηφιακό, μπορεί να είναι ενεργειακό σε σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά σε παραδοσιακά ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα. Στην Ελλάδα ποτέ δεν είχαμε σωστή οργάνωση των αγορών, αλλά πιστεύω ότι με την κρίση τα πράγματα πήγαν χειρότερα. Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Ε, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα τρόφιμα και βασικά είδη κατανάλωσης, ε, δηλαδή είναι ακριβότερα από τον ευρωπαϊκό Μέσο όρο βάσει στατιστικών στοιχείων, τη στιγμή που κατά τη διάρκεια της κρίσης το κατακεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Ελλάδα έπεσε από το 94% της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω στο 70%. Επομένως αυτή η ακρίβεια που μπορεί να έχει σχέση και με τη δομή της αγοράς γίνεται σκληρή και άδικη σε συνθήκες πτώσης του εισοδήματος. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι τα δημόσια έργα και οι κατασκευαστικές εταιρείε. Υπάρχουν ένα σωρό εκθέσεις, για παράδειγμα της Τράπεζας της Ελλάδος, που βλέπουν ότι κοστίζουν τα δημόσια έργα στην Ελλάδα περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε να κοστίζουν, ίσως γιατί η αγορά δεν λειτουργεί σωστά. Αυτός ο προβληματισμός με τις κατασκευαστικές εταιρείες και τα δημόσια έργα πήρε και μια δραματική διάσταση με τα γεγονότα στη Βουλγαρία. Πρώτον, το αυτοκινητιστικό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε 18 ανθρώπους, ίσως κατά εκτίμηση λόγω του κακού οδοστρώματος παρά το γεγονός ότι ο νέος εθνικός δρόμος ήταν, είχε χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά έχουμε και την δολοφονία της δημοσιογράφου Μαρίνοβα που έψαχνε αυτά τα ζητήματα. Ε, θέλω να ρωτήσω, με αυτά τα θέματα, δηλαδή τρόφιμα στην Ελλάδα ή κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία και κόστος δημόσιων έργων, ασχολείστε ή επειδή πρέπει οπωσδήποτε να έχετε μία ιεράρχηση, πάτε στα πολύ μεγάλα και αφήνεται κάποια άλλα που και αυτά όμως έχουν τη σημασία τους. Ευχαριστώ. Oh, but you are so very right. Ε, έχετε απόλυτα δίκιο ότι έχουν τη σημασία τους και αυτά τα θέματα, γιατί αυτά είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε σχεδιάσει ένα μοντέλο που μπορεί να εμπνεύσει και άλλους. Τι έχουμε, έχουμε εθνικές αρχές ανταγωνισμού που επιβάλλουν και αυτές ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού εντός της εθνικής αγοράς κάθε φορά. Και κάτι που έκανε ο προκάτοχός μου ήταν να χαρτογραφήσει όλες τις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών ανταγωνισμού. και βεβαίω σε πολύ στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Καμιά φορά οι εθνικέ αρχέ ανταγωνισμού χρειάζονται περισσότερη ανεξαρτησία. Και αυτό είναι ακριβώ εκείνο που συμπεριλαμβάνει η πρόταση που και επίσημα ελπίζω να εγκρίνουμε πάρα πολύ σύντομα. Και τα κράτη-μέλη και η Ελλάδα ελπίζω να τα υλοποιήσουν όλα αυτά. Γιατί το θέμα της ανεξαρτησίας, γιατί έχει σημασία ότι οι αρχές ανταγωνισμού δεν φέρνουν πάντα καλές ειδήσει στις κυβερνήσεις. Καμιά φορά κάνουν ανάλυση στην αγορά και βρίσκουν ότι κάποια αγορά δεν είναι καλά οργανωμένη. Δεν εντοπίζουν μόνο με μονομένες περιπτώσεις, αλλά κάνουν και κλαδικές έρευνες για να δουν πώς λειτουργεί ένας κλάδος και πώς είναι οργανωμένος, πώς έχει ρυθμιστεί. Και ελπίζω η πρόταση στην οποία έχουμε καταλήξει από κοινού, σε στενή συνεργασία θα είναι μεγαλύτερη αλεξαρτησία, περισσότερη πόλη, καλύτερα εργαλεία και υψηλότερα πρόστιμα φυσικά. Για να υπάρχει ένα μεγάλο αντικίνητρο και οι εταιρείε να μην ε, μπαίνουν σε συμπεριφορές κατά του καταναλωτού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, ε, το 85% των αποφάσεων που παίρνονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, Ανταγωνισμού λαμβάνονται από τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού. Πολύ πρόσφατα ήμουν στην Αθήνα και είχα τη χαρά να συναντηθώ ε, με τους ομολόγους μου της Αρχής Ανταγωνισμού στην Ελλάδα που είναι πάρα πολύ προσιλωμένοι στο έργο τους αυτό και ε, στο να υπηρετούν ε, τους Έλληνες καταναλωτές. Και στην Ελλάδα λοιπόν και στη χώρα μου και σε άλλες χώρες οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού ε, έχουν τη σημασία τους και σημασία έχει να απευθύνονται σε αυτές οι πολίτες και οι καταναλωτές όταν βλέπουν ότι κάτι πάει στραβά. Ότι υπάρχει κίνδυνος να έχουμε ένα καρτέλ στις κατασκευαστικές εταιρείες ή στην καθημερινή λιανική αγορά τροφίμων. Γιατί όπως και εμείς συνεργαζόμαστε ε, συνεχώς με την αγορά, το πράττουν και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού αυτό. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Ενίνα Αγγίλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Καλώς ήρθατε. Δύο θέματα έχω να θέσω. Πρώτα απ' όλα για το Brexit. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξασφαλίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υπονομεύσει τι 27 ε, χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον τη συμφωνία. Πολλά κράτη-μέλη ταυτόχρονα ανταγωνίζονται μεταξύ του για να προσελκύσουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν έδρα στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλε επιχειρήσει. ο διάφορου επιχειρηματικού λόγου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προτιμούν ένα κράτο μέλο από ένα άλλο. Πράγματι, η παίζει ένα σημαντικό ρόλο να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει ρυθμιστικό ανταγωνισμός στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά δεν έχω πιστεί ότι μπορεί να ακολουθήσει ολιστική προσέγγιση από αυτού. Από πλευρά ανταγωνισμού, πώς εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν ε, ισότιμοι όροι. Προβληματίζεστε για τα κριτήρια που χρησιμοποιούν αυτές οι αποφάσεις για εγκατάσταση. Τι προσπαθώ να πω. Πόσο σίγουροι είσαστε ότι τα κράτη-μέλη δεν προσελκύουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλου είδους ιδρύματα με ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση ή με άλλα κίνητρα. Δεύτερο, αφορά την αλλαγή του κλίματος. Πρόσφατα σε αρκετέ ομιλίε μιλήσατε ότι χρειαζόμαστε πιο βιώσιμη οικονομία. Η αλλαγή του κλίματο πράγματι είναι πολύ επικαιρό θέμα. Αυτή την εβδομάδα ε, με την έκθεση των ΗΕ που λέει ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προσπάθεια και τεράστιες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε και παρά όλη την νομοθεσία που έχει θετήσει το Κοινοβούλιο επί σειρά ετών, δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με κανόνες περί ανταγωνισμού να κινηθεί κατά των κακών ε, πρακτικών που ακολουθούνται για τη μετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Το συγκρίνω αυτό με το έργο που έχει γίνει όσον αφορά τη φοροδιαφυγή. Διότι μόνο όταν ξεκινήσατε να εξετάσετε τα θέματα Παναμά και τα tax rulings ότι αυτό έγινε πιο επίκαιρο θέμα, πιο σημαντικό θέμα και κινήθηκαν και τα κράτη-μέλη και προσελκύστηκε και η προσοχή του κοινού. Μήπω έχουμε αντίστοιχη εξέλιξη για την ε, πολιτική για το κλίμα, δοθέντως ότι οι κανονισμοί για το ETS ε, δημιουργήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δημιουργεί πρώτη του κανόνε, βλέποντα μετά το τοπίο το ενεργειακό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυριαρχεί εκεί πέρα κυριαρχείται από ελάχιστους φορείς και αντιμετωπίζει όλο και αυξανόμενο κόστος ενεργειακό Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως υπάρχει κάτι που μπορεί να εξεταστεί εκεί πέρα. Um, Κατανοώ αυτό που είπατε ότι οι εταιρείε πρέπει να υφθούν μια ολιστική προσέγγιση, έστω και αν δρούν τοπικά. και θα μπορούσαμε να δίνουμε κάποια φορολογικά κίνητρα, αλλά αυτό πρέπει να αφορά πρόσβαση σε ειδικευμένου ανθρώπου, υποδομέ, την εγκύτητα στην αξία παράγουν άλλε επιχειρήσει, στην περιοχή κλπ. Συμμετοχή στην αλυσίδα αξία. Αυτό είναι κατανοητό. Πάντω δεν έχουμε δει ακόμη τέτοιου είδου φορολογικά κίνητρα οποία να είναι πηγή ανησυχιών. Η συνθήκη πάντως δημιουργεί, προσφέρει τη δυνατότητα φορολογικού ανταγωνισμού και βλέπουμε διάφορες κινήσεις, πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. Ε, αυτό κάποια στιγμή πήραμε απόφαση να το αφήσουμε στη συνθήκη, όμως αντιμετωπίζουμε επιθετικά πραγματικές κρατικέ ενισχύσει. Τα προσέχουμε όλα αυτά πάντω να το ξέρετε. Επίση, πρόσφατα πήραμε μια απόφαση. Ε, ξέρετε, έχει σχέση με την Jaguar και την ε, απόφασή τη να δημιουργήσει εργοστάσιο στη Σλοβακία. Μεγάλη επένδυση τη Jaguar, πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Η ενίσχυση είναι περίπου 125 εκατομμύρια. Το ερώτημα είναι ποιο θα ήταν η εναλλακτική λύση για την συγκεκριμένη εταιρεία. Θα ήταν να πάει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ μπορούμε να δικαιολογήσουμε την ενίσχυση για μετεγκατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι εκτός. Οπότε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να τύχει έγκριση με τέτοια ενίσχυση. αλλά δεν μπορώ να φανταστώ κάτι παρόμοιο στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Τώρα για τη μεταβολή του κλίματος και ασχολούμαστε με το θέμα, το ξέρετε. Το θέμα είναι ότι ο τρόπο παραγωγής και χρήσης ενέργειας αλλάζει. Κάθε φορά που συμβαίνει μια εξέλιξη, το ενεργειακό μας σύστημα συνειδητοποιεί κάποια άλλη αδυναμία. Το θέμα είναι να έχουμε εφεδρείε, ξέρετε, στην παροχή ενέργεια Αυτό είναι το υπερθυμόν ένα ζήτημα. Αυτό το, το κάνουν τα κράτη-μέλη και είναι πολύ προσεκτικά να μην στρεβλώσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Πολλές φορές ε, αυτό είναι κακό για τις ανανεώσιμες πηγές. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε πληθυρικούς διαχωνισμούς ή μάλλον πληθυρικούς διαγωνισμούς γιατί τις ενισχύσεις. Μετά έχουμε αιωλικά πάρκα, τα οποία δημιουργούνται με μηδέν ενίσχυση. Και αυτό είναι καλό εν ώψη της μεταβολής του κλίματος. Το σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων, όπως πήρε και εσείς, ε, αλλάζει, μεταρρυθμίζεται. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε και τους δικούς μας εθνικούς κανόνες για το ETS, το σύστημα αυτό. θα μεσολαβήσει δημοσία διαβούλευση, η οποία θα ξεκινήσει μάλιστα και σύντομα ακριβώς για να εξασφαλίσουμε υποστήριξη για αυτήν την νομοθεσία και μετά να την εφαρμόσουμε βεβαίω. Άρα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε αυτόν τον τομέα και για τους κανόνες κρατικής ενίσχυσης. Δηλαδή οι ενισχύσεις αυτές είναι για καλό. Γιατί μερικά κράτη-μέλη χρειάζονται αυτά τα συστήματα εφεδρείας όταν περνούν σταδιακά προς την υδροελεκτρική, ηλιακή ή αιωλική ενέργεια. Ευχαριστώ, Μάρκος Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε, και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά είχαν έρθει κάτι εφοριακοί από την εκλογική μου περιφέρεια, ομάδα επισκεπτών, και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, να δούμε τι κάνουμε στα φορολογικά και κατάφερα πολύ ωραία να τους περιγράψω την πολιτική σας για τις κρατικές ενισχύσεις. Έρχομαι στο ψηφιακό κόσμο. Λέτε ότι έχετε τα εργαλεία ε, για να το αντιμετωπίσετε, αλλά η υπόθεση Google έχει αποδείξει το αντίθετο, γιατί η διαδικασία και ε, η διάρκεια της διαδικασίας είναι αιωνιότητα για την ψηφιακή εποχή. Είναι απαράδεκτος χρόνος. Πολλές εταιρείες να βάγισαν γιατί δεν είχαν καθόλου την ευκαιρία να τα βγάλουν πέρα απέναντι στη δεσπόζουσα θέση της Google, ούτε καν να αναπτυχθούν, ούτε καν να συσταθούν. Πρόσφατα έμαθα για δύο περιπτώσεις και θέλω να ρωτήσω αν είναι δεσπόζουσα θέση ή όχι. Στις υπηρεσίες πληρωμών, η Apple για παράδειγμα, έχει μια εφαρμογή που λέγεται NFC και ε, αποκλείονται ε, από αυτές τις ε, πληρωμές και το ίδιο ισχύει και με τη τεχνολογία Amazon που επιτρέπει μόνο το δικό του σύστημα πληρωμών ε, και όποιο άλλο θέλει να επιλέξει ένα διαφορετικό δρόμο δεν μπορεί να παραγγείλει κάτι από το Amazon. Αυτό είναι δεσπόζουσα θέση. Τι ε, επικρατεί εκεί στην αγορά και μέχρι να τα ελέγξετε όλα αυτά, τα μονοπόλια αυτά θα έχουν ευρεωθεί. Δεν μπορούμε να έχουμε πιο ταχεία δράση και να ε, επιβάλλουμε στις εταιρείες να δέχονται και άλλα συστήματα πληρωμών για να υπάρχει ε, ακριβώς ένας θεμητός ανταγωνισμός. Έχουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο να εφαρμόζονται και σωστά όλα αυτά. No, not at all. Είναι τα ερωτήματα που έχουμε και εμείς. Πώς θα επιταχύνουμε το έργο μας. σε αποδεκτό χρόνο. Να γίνουν αυτά σε αποδεκτό χρόνο. Υπάρχει και ένα όριο. Υπάρχει μια ιδιωτική συμμετρία εδώ. Κάποιος θέλει πέντε λεπτά για να διαρρήξει το σπίτι σα, να κλέψει τα... τη μαλφή και να φύγει. Ε, και μετά τρέχει από πίσω η αστυνομία και η δικαιοσύνη και από αυτό μπορεί να πάρει εβδομάδε για να βρουν τον α, ε, υπέτειο κλπ και μετά μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αποδείξει το δικαστήριο ότι ήταν πραγματι ένοχος. Αυτή η θεμελιώδης ασυμμετρία προκύπτει από το απλό γεγονό ότι ο κλέφτης, ο διαρρήκτης εν προκειμένου, δεν δεσμεύεται από το κράτος δικαίου, το οποίο είναι για μας αρχή. Άρα, αλλά συμφωνούμε όλοι μας ότι δεν θα παραβούμε ποτέ τους κανόνες της δικονομίας. Τώρα, μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να επιταχυνθεί η σχετική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Ε, προσπαθούμε να δούμε λοιπόν αν και στα δικά μας ζητήματα μπορούμε να κάνουμε κάτι προσωρινά. Γιατί η δίκη θα κρατήσει χρόνια, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Μπορεί όμως, να λάβει κανείς προσωρινά μέτρα, κατεπήγοντα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ακόμα και αυτά τα μέτρα όμως δεν θα είναι επαρκή. Γι' αυτό και ζήτησε από τους τρεις συμβούλους που προανέφερα να μας βοηθήσουν. Εν μεταξύ προσπαθούμε και εμείς να ψηφιοποιηθούμε και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν, για παράδειγμα, κατεβάσουμε δεδομένα μαζικά 7.000 ε, έγγραφα μια εταιρεία να κατεβάσουν στους υπολογιστέ μας Πρέπει να τα ανοίξουμε, τα διαβάσουμε και να δούμε αν υπάρχει τεκμήριο απόδειξη κάποιες παρανομίας. Για να γίνει αυτό, ας πούμε για να ταξινομήσουμε ακόμη τα 7.007 έγγραφα, χρειαζόμαστε ψηφιακή τεχνολογία. Αλλιώς δεν έχεις πρόσβαση στα έγγραφα. Και αν ε, δεν υπάρχει και τάξη σε όλο αυτό το υλικό, τότε χαθήκαμε. Και μιλώ μόνο για την διοικητική πτυχή της έτσι. Εδώ μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο. Να διευκολύνουμε λοιπόν την πρόσβαση στα έγγραφα, στα στοιχεία, ειδικά όταν οι φάκελοι, το πρωτογενές υλικό βρίσκεται σε μια αρχική κατάσταση. Όλα αυτά παίρνουν καμιά φορά εβδομάδες. Λοιπόν, αυτό δεν λέω, δεν λέω ότι σημαίνει ότι δεν πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα τη νομοθεσία. Όχι, αλλά πάντα υπάρχουν τρόποι να κάνουμε τη δουλειά μα καλύτερα και πιο γρήγορα. Για τα δύο παραδείγματα που αναφέρατε, ε, να ξέρετε ότι τα παρακολουθούμε και τα δύο. Το θέμα είναι το εξή. Η δρανοποίηση άλλων ε, υπηρεσιών προκαλεί το εξή πρόβλημα. Το θέμα είναι καταρχήν αν είναι μια δεσπόζουσα θέση ή όχι. Αν δεν είναι, ο καταναλωτής ενοχλείται, αλλά δεν υπάρχει παρανομία. Αν είσαι σε δεσπόζουσα θέση, από την άλλη μεριά, μπορείς να κάνεις πράγματα νόμιμα, το οποίο ενοχλούν, τα οποία δεν επιτρέπονται, επειδή είσαι σε δεσπόζουσα θέση. Επιτρέπονται όμω για μια μη δεσπόζουσα επιχείρηση. Τα παρακολουθούμε πάντω αυτά, παρακολουθούμε το θέμα των ε, στοιχείων όπω ξέρετε. Ψάχνουμε και την Amazon πώ αξιοποιεί τα στοιχεία. Τα στοιχεία μάλιστα των ε, εμπόρων, των μικρών επιχειρήσεων που φιλοξενεί η Amazon, που πολλούν δηλαδή αυτοί μέσω τη Amazon και το πώς επιτρέπει και πώς χειρίζεται η Amazon τις περιπτώσεις τους. Ε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορώ να σα δώσω επιπλέον. Πολ Τάγκ, πρόεδρε. Είναι πολύ ε, μεγάλος ο πειρασμός να, να κυριαρχήσει κανείς την αγορά. Εγώ θα ασχοληθώ με ένα άλλο θέμα. Επιχειρήσεις που έχουν δύο έδρες. Ολλανδική και Βρετανική. Unilever και Shell πίεζαν για κατάργηση αυτές οι εταιρείε. Λοιπόν, ένα δημιονέκτημα αυτών των εδρών είναι η φορολόγηση και ζητούσαν κατάργηση του οριστικού φόρου, του μόνιμου φόρου που είναι βάρος για τους Βρετανούς μετόχους. Εμποδίζουν αυτοί οι φόροι τις εταιρείε. Και είχαμε και tax ruling στην περίπτωση του, τη Shell το 2005. Φορολογικός εμπειρογνώμων μελέτησε την υπόθεση και συνεπέρανε ότι πιθανότατα είναι κατά του Ολλανδικού νόμου, της Ολλανδικής νομοθεσίας. 7,5 δις αφορούσε αυτό, αυτή η απόφαση εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτές οι εταιρείε δημιουργείται πρόβλημα που έχουν δύο έδρες και που ασκούν πιέσεις για tax ruling και ειδική αντιμετώπιση. Και την υπόθεση Shell του 2005 που ε, κατήγγειλε ο Γιάνν Βενστρέκ, ο ειδικό ε, για θέματα εφορία, ε, εφορίας. Ε, ναι, γνωρίζουμε. Εσείς το θέσατε προηγουμένω, λέει Επίτροπος. Υπήρξε και αρκετή κάλυψη από τα ΜΜΕ. Ναι, δώσαμε συνέχεια και δίνουμε συνέχεια στις πληροφορίε που δίδονται και να έχει τι καλές πληροφορίε με τα χαρά να τις λάβουμε υπόψη. Συνέχεια τι εννοείται. Ότι θα εξετάσετε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Απάντηση ναι, ήδη το κάνουμε. Όπως σας είπα, το συζητήσαμε και πριν το θέμα αυτό στην υπόθεση. Παρακολουθούσαμε επίσης και τις αναφορές στον τύπο. Δεν έχουμε συγκεκριμένη δικογραφή υπόθεση του ΣΥΠΗΝ. Θέλουμε να καταλάβουμε όμως ενδελεχώς την υπόθεση, να δούμε εάν υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει πραγματικά μια υπόθεση που πρέπει να εξηχνιαστεί. Βέρνερ Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Δύο ερωτήσεις έχω πρώτη ερώτηση. Σε σχέση με αυτό που ρώτησε η κυρία Μπερές, φορολογικός ανταγωνισμός. Εσείς γράψατε ιστορία με την υπόθεση Apple στην Ιρλανδία. Και ε, τέλη Σεπτεμβρίου είχε εξαγγελθεί ότι θα καταβληθούν οι πληρωμές. Καταβλήθηκαν. Τι γίνεται και, και πριν, την, ε, πριν η υπόθεση θα μπορέσετε να έχετε δημιουργήσει τελεσμένα. Και συζητήσαμε επίσης και την υπόθεση της Μαδέρας. Αντίστοιχα συμβαίνουν και στη Μάλτα. Στις συνθήκες προσχώρησης λέει ότι εξωτερικές εταιρείες ε, πληρώνουν 5%, οι ντόπιες 30%, 25% διαφορά. Ε, αυτό όταν είναι μεταβατικό έχει καλός, όχι μόνιμο όμως όπως συμβαίνει στη Μαδέρα δεν μπορεί να είναι σε μειονεκτική θέση εγχώριες εταιρείε στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Θα κάνετε τίποτα. Και η τρίτη υπόθεση είναι οι άδειε στις κάτω χώρες που είναι ε, πάνω από ε, αθέμητος ανταγωνισμός γιατί τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι άδειε δεν φορολογούνται στην Ολλανδία και πάνε όλες οι εταιρείε αυτές και εγκαθίστανται εκεί θα κάνετε τίποτα, γιατί επειδή υπάρχει ομοφωνία στα φορολογικά, είστε ε, οι μόνοι που μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δικαστήρια. Ε, εγώ σας θαυμάζω για τη δουλειά που κάνετε. Ε, αλλά και στην ίδια σας την πατρίδα υπήρξε ένα σκάνδαλο ξεπλήματος με τη μεγαλύτερη ιδανική τράπεζα. Είστε πάντως σε καλό δρόμο. Και το επόμενο θέμα που θέλω να ρωτήσω, το τρίτο, έχει να κάνει με τις συμβάσεις ανάμεσα στους ε, αντιπροσώπους διαφόρων αυτοκινητοβιομηχανιών που ε, ε, χαίρουν διαφόρων εξαιρέσεων ομαδικών. Μου απαντήσατε το καλοκαίρι σε μια επιστολή ότι τα μελετάτε. Ενέχονται και δύο γερμανικές εταιρείες. Η Volkswagen για τους αντιπροσώπους και η BMW είναι η δεύτερη περίπτωση, την οποία εγώ γνωρίζω σε λεπτομέρειες για κάποιες ατέλειες στο δίκτυο αντιπροσώπων τους. Ναι, πράγματι, οι πληροφορίες για την Apple που κατέβαλε τους μη καταφληθέντες φόρους είναι ορθοί, πλήρωσαν μαζί με τους τόκους τους φόρους 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ έδωσε η Apple σε ειδικό ε, ταμείο, σε ειδικό λογαριασμό και έτσι σταματάει η δικαστική υπόθεση διότι προσφύγαμε στο δικαστήριο διότι δεν είχε καταβληθεί πληρωμή. Τώρα όχι μόνο δόθηκε προκαταβολή αλλά καλύφθηκε πλήρως. Οπότε σταματήσει η δικαστική αγωγή κατά της Ιρλανδίας γι' αυτό. Για τη Μαδέρα εξετάζουμε κατά πόσο αυτά τα ειδικά πλαίσια για τη Μαδέρα χρησιμοποιήθηκαν σωστά για το σωστό σκοπό. Διότι η Μαδέρα έχει και κάποια προβλήματα, δεν είναι στην υπηρετική Ευρώπη, οπότε επιτρέπεται ειδική κάλυψη, ειδικά μέτρα για τη Μαδέρα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και για ενίσχυση δραστηριότητα. Και αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό εξετάζουμε τώρα. Και βέβαια ε, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την έρευνα το το δυνατό. Το θέμα, το ερώτημα της Μάλτας, μπορείτε να το επαναλάβετε παρακαλώ. Η Μάλτα ε, φορολογεί διαφορετικά τους ξένους επενδυτές από ό,τι τους εγχώριους. Το διαπραγματεύθηκε στην ένταξή της ως μόνιμη λύση, αλλά κατά την άποψή μου μετά από μία δεκαετία θα έπρεπε να έχει τερματιστεί αυτή η ιστορία. Ε, we have, uh, this... Απάντηση. Έχουμε ειδικέ διατάξεις όσον αφορά τις υφιστάμενες ενισχύσεις. Αυτό ισχύει για κάθε κράτος μέλος όταν γίνεται η ένταξη στην Ένωση. Υπάρχουν ειδικέ διατάξεις για υφιστάμενες ενισχύσεις και μπορούμε να το εξετάσουμε αν δούμε ότι έχει εκπνεύσει το διαπραγματευτικό πρωτόκολλο. Μέχρι τώρα για το θέμα της Μάλτας δεν έχουμε θέσει ερωτήματα, αλλά θα το ερευνήσω και θα επανέλθω για την Ολλανδία και κατά πόσο ε, ε, τι γίνεται με τη φορολόγηση των πνευματικών δικαιωμάτων, η αξία που δημιουργείται πνευματικά δικαιώματα αν φορολογείται. Αυτό το ΩΣΑ το εξέτασε. Τι βρήκαν στον ΩΣΑ. Μία διευθέτηση όπου θες να προωθήσεις έρευνα και ανάπτυξη και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται. Αυτό είναι θεμητό. Α, επιτόπου. Αν επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη, για την έρευνα και ανάπτυξη προκύπτει ένα πνευματικό δικαίωμα, μια βρεσιτεχνία, ε, εκεί καλύπτει με ειδικέ διατάξει τα έσοδα προέρχονται από το πνευματικό δικαίωμα. Εάν μπορεί να προέρχεται από οδήποτε πνευματικό δικαίωμα και προκύπτει εισόδημα που δεν φορολογείται από το πνευματικό δικαίωμα, αυτό θέλουμε, από αυτό θέλουμε να απαλλαγούμε. Δεν θέμα φορολογικό, είναι θέμα του Πιέρ Μοσκοβισή. Και ήδη έχει θεσπίσει νομοθεσία το Συμβούλιο για να γίνει δέουσα αλλαγή. Αυτό που αποκαλεί ο ΩΣΑ, αυτό που θεωρεί ο ΩΣΑ νόμιμο, διότι προωθεί την έρευνα και ανάπτυξη επιτόπου, ευρωπαϊκή επένδυση επιτόπου για, σε συγκεκριμένη χώρα για έρευνα και ανάπτυξη, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ε, το πνευματικό δικαίωμα την ευρεσιτεχνία για να μην φορολογήσει. Για τα πορίσματα στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα καρτέλ, δεν έχουμε ακόμα επιβεβαιώσει τις υπόνοιές μας, αλλά έχουμε σαφή, σαφή συγγνώμη στόχευση τώρα για την υπόθεση. Είναι καλό αν η αυτοκινητοβιομηχανία συνεργάζεται για θέματα ασφαλεία και μέτρα ασφαλεία. Αυτό ωφελεί του καταναλωτέ. Ε, και στο μέλλον θα δούμε ότι θα συνεργάζονται οι εταιρείε αυτοκινήτων, κατασκευή αυτοκινήτων για το πώ θα χρησιμοποιούν τι μπαταρίε με έναν τρόπο που να μπορούν να ανακυκλώνονται. Οπότε υπάρχουν διάφορε περιστάσει όπου συγκεκριμένα λέμε εδώ η συνεργασία είναι θεμητή. Τώρα για την έρευνα για καρτέλ στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ποια είναι η ανησυχία μας. Ότι υπάρχει καρτέλ για τη μη χρήση των βέλτιστων τεχνολογιών για πιο καθαρές εκπομπές και για τα αυτοκίνητα με ε, βενζίνη και με ντίζελοκινητήρες. Δεν είδαμε να υπάρχει σχέση μεταξύ του σκανδάλου εκπομπών και του καρτέλ που ερευνούμε τώρα. Το σκάνδαλο των εκπομπών ακόμα εξετάζεται από ομάδα συναδέλφων μου, με τον κύριο Κατάινεν σαν επικεφαλής. Ο πρόεδρος, ε, τελειώνει ο χρόνος μας. Ε, ε Λάγκεν, ε, μια σύντομη ερώτηση μόνο. Για ε, τον κανονισμό εξαίρεσης κάποιων ομίλων που είναι μέχρι το 2023. Υπάρχουν κάποια εργοστάσια αυτοκινήτων που έχουν μικρομεσαίους αντιπροσώπους οι ε, ε, ε, πολιτές αυτοκινήτων. Αυτή τη νομοθεσία την περιφρονεί και την παραβιάζει η Volkswagen. Ε, κοιτάξτε, το δούμε διμερώς αυτό. Είναι δευτερεύον σε σχέση με αυτό που έλεγα προηγουμένως για το καρτέλ στην αυτοκινητοβιομηχανία. Good. Μάλιστα. σου έχω δώσει παραπάνω χρόνο και μη διαμαρτυρηθείς αν θα δώσω και σε άλλους συναδέλφους. Ο Ραμόν Χάουρεγγι. Δεν θέλω το λόγο. Yes. Okay. No, you were... Χωρίς μικρόφωνο, κύριος ε, ε, Είχαμε το όνομά σας στον κατάλογο, δεν θέλετε το λόγο. Ωραία. Κάτσε διάει έχουμε. Ε, όχι. Ε, ε ολοκληρώνουμε εδώ. Ακριβώς την ώρα μας. This, uh, excellent... Αυτή την εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων. Το διαρθρωμένο διάλογο με την κυρία Βεστάγκερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζεται φυσικά ο διάλογος και προσβλέπουμε σε αυτό πολλά τα θέματα. Ε, θα χρειαστεί και συνέχεια να δοθεί σε όλα τα επίπεδα. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε αγαστή συνεργασία μαζί σας. Και να πάτε στο καλό και ό,τι επιθυμείτε. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, σημείο 17, επιβαρύνσεις της διασυνοριακής πληρωμές στην Ένωση και τέλη μεριτροπών συναλλάγματος. Έχουμε 104 τροπολογίες, 14 από του σχεδίου έκθεσης, οπότε δίνω τον λόγο για τέσσερα λεπτά στην εισηγητρία και μετά έχουμε του Σκιώδη και catch Αν προλαβαίνουμε βεβαίω εντό των 30 λεπτών. Εύα Μάιντελ από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήμουν σε διάλογο με του πολίτε αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ θερμά τους Σκιώδη και τους αδελφού τη ΕΚΟΝ για τις επικοδομητικές προτάσεις που υπέβαλαν εν ώψη τροπολογιών. Έχουμε την ευκαιρία να νομοθετήσουμε ώστε να φέρουμε πιο κοντά τους πολίτες και να λύσουμε μερικά από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν μεταφέρουν χρήματα από τη μία χώρα στην άλλη. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να δείξουμε στους άπιστους θωμάδες ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα προχωράει και ότι βελτιώνει εν τέλει τη ζωή των πολιτών εξοικονομώντας και χρήματα στο πλαίσιο της εκπόνησης της γνωμοδότησης ε, θα συμβάλλω και εγώ ελπίζω στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Χαίρομαι ε, διότι πολλές από τις προτάσεις είναι φιλόδοξες, διευρύνουν το πεδίο εφαρμογή των διασυνοριακών μεταφορών. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο κατηγορίες προβλημάτων. Έχουμε τις υπηρεσίε πληρωμών που είναι κατακαιρματισμένες αλλά ζούμε σε μια ένωση και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ε, άρα λοιπόν έχουμε ανθρώπους που στέλνουν χρήματα από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτές οι μεταφορές πρέπει να επιβαρύνονται με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, είτε είναι πρόκειται για ευρώ είτε για άλλο νόμισμα. Επίσης, οι πάροχοι αυτών των συστημάτων πληρωμών ε, επεξεργάζονται ήδη με αρκετή ταχύτητα τέτοιου είδου μεταφορέ. Το επιχείρημα όμω ότι δεν υπάρχει κεντρική Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Εκαθάρισης ε, δεν είναι πιστικό επιχείρημα όταν η τεχνολογία επιτρέπει την ταχύτατη λειτουργία και τις ελαγές ε, στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις αυτές να καινοτομήσουν για το καλό των οικονομιών μας. Έτσι λοιπόν υπάρχει υπηρεσιών πληρωμών και οι τράπεζες πρέπει να βρουν λύσεις. Νομοθετούμε λοιπόν για να μειωθούν αυτές οι επιβαρύνσεις. Φυσικά αυτό δεν πρέπει να αντισταθμιστεί με αυξήσεις σε άλλους τομείς, για άλλες υπηρεσίες. Εδώ θα επαγρυπνήσουμε. Σε επίπεδο POS, σε επίπεδο ATM. Κύριε Λουτβίνσκι Βίχσεν ε, και άλλοι συναδελφοί έχουν υποβάλει σχετικέ τροπολογίε. Χρειαζόμαστε επίση νομική ασφάλεια και ευκολότερη συμμόρφωση. Το θέμα είναι ότι κανεί καταναλωτή δεν κουβαλάει μαζί του κομπιουτεράκι όταν αποσύρει χρήματα από ένα ATM ή όταν ψωνίζει. Οπότε πρέπει το κόστος αυτό να είναι διαφανές. Δεν εμφανίζεται σαφέστατα και στα δύο νομίσματα όταν έχουμε να κάνουμε μετατροπή για να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ο καταναλωτή. Και οι δύο λοιπόν εναλλακτικέ λύσει πρέπει να παρουσιάζονται ταυτόχρονα και όχι παραπληνητικά σε διαφορετικό χρόνο. Για να μπορέσει, όπω είπαμε, να πάρει τη σωστή απόφαση ε, ο καταναλωτή Κάρα, Ζεντερμάγερ, Γέζεκ και όσο υπέβαλαν επίση ε, τροπολογίε και απαντώ, άκουσα ένα επιχείρημα από καταναλωτέ και οργανώσει του το λέει και ο κ. Λουτβίχσον στην ε, τροπολογία του 199, αφορά την ε, παροχη δικαιωματο δικαιώματος opt-in, opt-out για τη μετατροπή ενό νομίσματος. Πρέπει οι καταναλωτέ να ξέρουν ότι έχουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία και βέβαιω να αποφασίζουν αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικό τρόπο πληρωμή. Οι απαιτήσει περί διαφάνεια είναι πολύ σημαντικέ θα το συζητήσουμε περαιτέρω με όλους σας πώς θα πετύχουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Εύα. Ο κ. Λούντβιχσον ε, για τρία λεπτά έχει το λόγο από τους ηγητές μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την Εύα Μάιντελ για την έξοχη συνεργασία μας μέχρι τώρα και πιστεύω ότι οι επικοδομητικές συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν. Και στην επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών παρουσίασα τροπολογίες. Σε αυτές τις τροπολογίες επικεντρώνομαι επί της σημασίας που έχει να καλύψουμε τα νομίσματα όλων των κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάσουμε τα πράγματα σαφέστατα για τους καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ ξεκάθαρα ποιες είναι οι ισοτιμίε που θα πρέπει να πληρώσουν ή να μην πληρώσουν. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουν υπόση ε, και το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτω ώστε να είναι αποτελεσματικότατο το σύστημα. Είναι σημαντικό να μειωθούν τα τέλη που αφορούν τις διασυνοριακές συναλλαγές σε όλα τα κράτη, ανεξάρτητα από το νόμισμα. Είναι σημαντικό να μειωθεί το κόστος για τι διασυνοριακές πληρωμέ σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα θέμα ισότητα. Διερωτώ λοιπόν. Από πού ξεκίνησε ο προβληματισμός και η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι προφανές ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής θεωρεί ότι τα τέλη, το κόστος πρέπει να μειώσει για όλους όσους είτε ζουν στην Ευρωζώνη είτε όχι. Είναι πολύ σημαντικό ε, να μπορέσουμε ε, να δημιουργήσουμε δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των ισοτιμιών των διαφόρων ε, νομισμάτων. Στους υπολογισμούς περί ισοτιμίας λαμβάνουμε υπόψη ότι κάτι είναι πιο ακριβό ή πολύ πιο ακριβό σε μια χώρα που χρησιμοποιεί ένα νόμισμα σε σχέση με κάποιο άλλο θα πρέπει ο καταναλωτής να μπορεί να ενημερώνεται για την τιμή των προϊόντων και να μπορεί να επιλέξει σε ποιο νόμισμα θα ε, καταβάλει την πληρωμή. Και είναι σημαντικό, αυτό. Ε, είναι δύσκολη υπολογισμή καμιά φορά για τον μέσο καταναλωτή όταν τον πιέζει ο χρόνος θέλει να αγοράσει κάτι. Γι' αυτό στην τροπολογία 102 προτείνω διάφορα μέτρα, μέτρα που θα επιτρέψουν καλύτερη συγκρισιμότητα μεταξύ των διαφόρων ισοτιμιών, μεταξύ των διαφόρων νομισμάτων, έτσι οι καταναλωτές μπορούν πιο εύκολα ε, να έχουν πρόσβαση σε διασυνορικές πληρωμές, να ξέρουν καλύτερα ποια ισοτιμία υπάρχει, τι πληρώνει ε, και ποιο ε, τέλος πρέπει να καταβάλει στον φορέα που κάνει την πληρωμή και το έμβασμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βρούμε μια λύση σε αυτό το θέμα, πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ συχνά ο, ο καταναλωτή δεν μπορεί να κάνει του δέοντε υπολογισμού. Αν θέλουμε ένα δυναμικό σύστημα, ε, θα πρέπει οι πληροφορίε να δίδονται σαφώ. Θα πρέπει ο καταναλωτή να είναι ενήμερο όσον αφορά το συνολικό κόστο που θα πρέπει να καλύψει, που θα πρέπει να πληρώσει και θα πρέπει να μπορεί να βρίσκει λύσεις άλλες αν το επιθυμεί. Αυτοί οι νέοι κανόνες περί διαφανείας θα πρέπει να τεθούν σε, σε ισχύ, να ισχύουν 12 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του κειμένου. Α, αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται και κατά την πληρωμή και κατά την ε, απόσυρση χρήματος. Ε, θα πρέπει όταν κάποιος χρησιμοποιεί ρευστό, ο καταναλωτής που θα χρησιμοποιήσει ρευστό να γνωρίζει ακριβώς ποιο είναι, ποια είναι η ισοτιμία και τι πρέπει να καταβάλει. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ έξι μήνες μετά τη θέση ισχύ του, κειμένου. Ε, διότι πρέπει να μπορούμε να λάβουμε υπόψη την καλύτερη δυνατή εφαρμογή. Είμαι πεπισμένο ότι θα συνεργαστούμε του επόμενου μήνε επικοδομητικά και τι επόμενε εβδομάδε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Είμαι σίγουρο ότι μαζί θα βρούμε μια έξοχη λύση προ όφελο του Ευρωπαίου καταναλωτού. Ο Από ε, του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ τη ΙΣΙΑ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, ευχαριστώ για τις συμβαστικές τροπολογίες, αλλά έχω μια σημαντική ερώτηση ως προς το περιεχόμενο στη συμβαστική πρόταση Α. Η κυρία εισηγήτρια ε, ξέρει πολύ καλά ότι και εμείς και οι σοσιαλιστές, αλλά και κάποια μέλη του ΕΛΚ ε, θέλουμε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή ε, κατάργησης ε, των τελών για τις διασυνοριακές πληρωμές σε όλα τα νομίσματα της Ένωσης, όχι μόνο στο ευρώ, για να τηρείται η αρχή της αμοιβαιότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού ε, για τον κλάδο των πληρωμών ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα τα νομίσματα είναι ισότιμα. Δυστυχώς όμως η συγκήτρια δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις μας στη συμβαστική α βλέπω ότι οι τράπεζες εκτός της Ευρωζώνης ουσιαστικά θα πρέπει ε, να επιβάλλουν τα δικά τους τέλη στις διασυνοριακές προμές και τα εμβάσματα σε όλα τα νομίσματα πλην του ευρώ. Ενώ εντός της Ευρωζώνης οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να κάνουν το ίδιο ε, για τα ίδια τέλη και για τις ίδιες διασυνοριακές πληρωμές ε, σε νομίσματα πλην ευρώ. Δεν ισχύουν λοιπόν τα ίδια ε, μέτρα και τα ίδια σταθμά εντός και εκτός της Ευρωζώνης. Ε, αυτό έχει ε, επιπτώσεις για τους καταναλωτές και για τους πελάτες και μας προβληματίζει. Θεωρούμε ότι το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που διαβάζουμε στο λεγόμενο συμβιβασμό. Παρακαλώ να επιδείξετε αλληλεγγύη και σε αυτό το τομέα και για τις ε, πληρωμές και υπάρχει ένα θέμα ισότητας των κρατών μελών εντός ή εκτός της Ευρωζώνης. Δεν μπορούν να υπονομεύονται τα άλλα νομίσματα πλην του ευρώ να θεωρούνται νομίσματα δεύτερης κατηγορίας ή χειρότερα νομίσματα από το ευρώ, εν πάση περιπτώσει. Άλλο θέμα είναι το κόστος των συναλλαγών. υπάρχει ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ε, ε, ε, μία άλλη τιμή που προτείνουν οι συναλλασσόμενοι για τη μετατροπή. Θα πρέπει να ισχύει πάντα η ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πάντα με μία αποποίηση ευθυνών που να λέει ότι όλα αυτά είναι ενδεικτικά και όχι οριστικά. Και τι γίνεται με τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει το ευρώ, θα είναι σε χειρότερη μοίρα. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι η τράπεζα αναφοράς. Για ποιο λόγο εμείς να υιοθετούμε το δικό τους ε, ε, επιτόκιο ή την ισοτιμία τους κάθε φορά. Τα πράγματα αυτά ε, δεν είναι δύσκολα. Γιατί πρέπει να τα περιπλέκουμε. Μπορούμε να δίνουμε την ισοτιμία συν τα τέλη που να είναι όμως συγκεκριμένα και σταθερά και να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει. Κάτι άλλο που χρειάζεται εξήγηση είναι μια μυστηριώδης έννοια που είναι η πραγματική ισοτιμία. Τι είναι αυτό. Ε, αυτό είναι για πληρωμές που δεν γίνονται εκείνη τη στιγμή αλλά σε διαφορετικό χρόνο. Έχω και άλλα να πω για το κείμενο, αλλά μάλλον θα τα υποβάλω γραπτός για να είμαι βέβαιος ότι θα το συζητήσουν οι σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Από τους φιλελευθέρους δεν βλέπω κανέναν, αν δεν απατώμε. Δεν είναι κανείς εδώ. Από τους πρασίνους, ο κύριος Ρέιμον αποσιάζει. Ο κύριος Βιέγας από την Γουέ. Ναι, αλλά είναι ο κύριος Γκίγκολτ εδώ από τους πρασίνους. Take please. Έχετε το λόγο, κύριε Γκίγκολτ. Πρόεδρε, εν συντομία, και επί της ουσίας των τροπολογιών για να μην μακρηγορώ. Υποστηρίζουμε όλες τις τροπολογίες που ζητούν περισσότερη προστασία για τους καταναλωτές. Διάφοροι συνάδελφοι υπέβαλαν τροπολογίες. Υποστηρίζουμε κυρίως τη θέση ότι πρέπει όχι μόνο να αυθυραμιστούν διάφορες επιβαρύνσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ε, αλλά να συμπεριλάβουμε αυτό και τις μετατροπές σε άλλα νομίσματα. Και συμφωνούμε και με τις 35, 36 και 37 και αυτές του Λουδίξον που έχουν στόχο πλήρη διαφάνεια και συγκρισιμότητα τιμών διαφόρων υπηρεσιών μετατροπής και πριν από την συναλλαγή ε, γιατί δεν έχει πολύ νόημα να το, το μαθαίνεις μετά, εκ των υστέρων. Το θέμα είναι να επιλέγεις γνωρίζοντα το κόστος κάθε μεθόδου πληρωμής. Και αυτό πρέπει να γίνεται την ώρα εκείνη που πληρώνεις, Αλλιώ δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα. Και το λέω αυτό, διότι αν και συμφωνούμε με μερικέ τροπολογίε του κ. Ζοκ, δεν συμφωνούμε με την 176, η οποία προβλέπει γι' αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα ότι διαφάνεια, ότι διαφάνεια μπορεί να παρέχεται εκ των υστέρων. Συγγνώμη, αλλά έτσι δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα. Επίσης, καλή ιδέα οι χρήστες να μπορούν να αποκλείουν την μερατροπή σε άλλο νόμισμα, όπως το οποίο είναι και η τροπολογία του Λουδίξον να αποκλείουν την μετατροπή σε άλλο νόμισμα. Δεν το Χούμπνερ και βέβαια ο κ. Φλουτφίξον έχουν υποβάλει μια άλλη τροπολογία. Ε, διαφωνούμε με αυτήν γιατί την είδαν πολλοί συναδελφοί και φαίνεται ότι προέκυψε από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε τεχνικό τουλάχιστον επίπεδο. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν θέλουμε ανώτατο όριο χρεώσεων για τη μεταβατική περίοδο. Αυτό δεν το θέλουν πολλοί συνάδελφοι. Δηλαδή δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ένα ανώτατο όριο χρεώσεων στη μεταβατική περίοδο. Εδώ δηλαδή τα παίρνουμε χοντρά από τους καταναλωτές και ξαφνικά μια πρόταση που λέει ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ανώτατο όριο χρεώσεων κατά τη διάρκεια τη μεταβατική περίοδου μέχρι ότου ισχύσουν οι κανόνες που προστατεύουν τη διαφάνεια. Ένα παράδειγμα. Για την μεταβατική περίοδο, ίσα χρειαζόμαστε αυτήν την, αυτό το ανώτατο όριο χρεώσεων και είναι κρίμα πραγματικά ότι οι συνάδελφοι που είναι υπέρ αυτής τη αρχή, εδώ έπεσαν σε μια νομικήστικη παγίδα δέχτηκαν το επιχείρημα ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μπορεί να πάρει τέτοιε αποφάσει. Υπάρχει νομική βάση λοιπόν για τέτοιο ανώτατο όριο χρεώσεων και η EBA θα το θεσπίσει αυτό επισήμω, γιατί και αυτοί πρέπει να υπερασπιστούν τους καταναλωτέ στο καταστατικό τους. Προβλέπετε αυτό. Και είναι γνωστό ε, ότι οι αναλυτικές μέθοδοι κοστίζουν για τους καταναλωτές περισσότερο. Αυτή η ληστεία πρέπει να τελειώσει. Και το λέω και προς τον εισηγητή. Θα ήθελα να κρατήσουμε το σχέδιο του RTS όπως το είχε ε, γράψει η Κομισιόν. Γιατί έτσι, γιατί αυτό είναι προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών. Πρόεδρος, ο κ. Βιέγας, από την Καλημέρα, θα μιλήσω πορτογαλικά, όπως συνήθως. Έχω κάποια σχόλια να κάνω. Διδάσκω οικονομικά και κανονικά αντιστοιχεί στο εμπόριο η διαμόρφωση των τιμών. Είναι από τους βασικούς κανόνες αγορές, της αγοράς. Λοιπόν, θα πρέπει να τίνουμε προς το μηδέν όσον αφορά το κόστος, ε, τα τέλη που πρέπει να καταβάλουμε. Γιατί δεν γίνεται αυτό, διότι δεν υπάρχει οικονομία της αγοράς ανταγωνιστική. Στην Πορτογαλία το τραπεζικό σύστημα ε, είναι μονοπολείται από διάφορα ε, ιδρύματα φορείς που χειραγωγούν τις τιμές και τα τέλη στην ε, Πορτογαλία έχουν φτάσει σε αστρονομικά επίπεδα αυτές τις φορές. Η ευθυγράμμιση των διεθνών συναλλαγών με τις εθνικές συναλλαγές από την άποψη των Πορτογάλων καταναλωτών δεν είναι κάτι θετικό, αντιθέτως μάλιστα. Θα πρέπει να καθορίσουμε ένα όριο, ένα μέγιστο για να σταματήσει αυτή η τάση Αύξηση τεράστιας ε, των διαφόρων τελών που καταβάλλονται στις πληρωμές. Με την περίοδο που ακολούθησε την κρίση κατέρευσαν τα επιτόκια και βλέπουμε αυτή την έκρηξη των διαφόρων ε, εισφορών, αυτών των τελών που επιβάλλουν οι τράπεζες εάν κανείς στείλει ένα έμβασμα στο διαδίκτυο, πληρώνει 1,5 ευρώ. 1,50 ευρώ 50 Οι τράπεζες μαζικά έχουν απολύσει προσωπικό και έχουν εισαγάγει τεχνολογικά μέτρα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί τελικά αυτά τα τέλη δεν μειώνονται προς το μηδέν όπως θα επέβαλε και ο νόμος της αγοράς όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς. Όσον αφορά τα ATM, τα αυτόματα μηχανήματα για το ρευστό και αυτό είναι ένα πρόβλημα, όπως και υπάρχει και πρόβλημα διαφάνειας όσον αφορά την α, απόσυση μετρητών σε ξένο νόμισμα. Εμείς είμαστε διστακτικοί. Έχουμε αμφιβολίες όσον αφορά τη δυνατότητα να μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα φάσμα επιλογών στους καταναλωτές σύντομα. Η κατάσταση είναι ανησυχητική. Όμως δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τι θέλει ο καταναλωτής. Θέλει τις καλύτερες δυνατές συναλλαγές με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Και οι πάνω σε αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει σταδιακά να τίνουν προς το μηδέν. Ο, ο πρόεδρος Κατσδιάη, αν δεν σας πειράζει να πω εγώ δύο λόγια. Πρώτα μιλάμε για έλεγχο των τιμών. Και ο έλεγχος των τιμών δεν είναι έτσι κάτι που το κάνουμε άσκοπα. Είναι επειδή δεν λειτουργεί καλά η αγορά. Το είπε ο κύριος Βιέγας. Τα ολιγοπόλια εκμεταλλεύονται τις πόσες θέσεις που έχουν. Βέβαια, έλεγχο των τιμών καμιά φορά σημαίνει ότι κοινωνικοποιούμε το κόστος και το μετακυλούμε σε άλλους πελάτες. Ε, η συγκήτρια σίγουρα θα βρει τη σωστή ισορροπία. Εύα, θέλεις να κλείσεις, να πεις δύο λόγια. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και πάλι. Όπως γνωρίζετε, ε, το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφιχτό. Οι συμβαστικές τροπολογίες έχουν κυκλοφορήσει. Ε, δεν ξέρουμε πότε θα συνεδριάσουν οι σκιώδεις συζητητές. Θα δούμε, θα το κανονίσουμε για τα σχόλια. Παρόλο που δεν θα συζητήσουμε σήμερα τις ε, συμβαστικές τροπολογίες, θέλω να απαντήσω σε κάποια σχόλια των σκιωδών εισηγητών, ιδιαίτερα του ΙΣΙΑΡ. θα πρέπει να διευκρινίσω ότι το κείμενο της συμβαστικής τροπολογίας ΑΕ ε, είναι πιο κοντά σε αυτό που ζητούν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες και το ECR, αν το συγκρίνουμε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εγώ ζήτησα να ευθυγραμμιστούν ε, ε, τα τέλη ε, όχι μόνο στις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ αλλά και σε εθνικά νομίσματα. Ας πούμε αν στέλνει από τη Βαρσοβία στις Βρυξέλλες σλότη, πολωνικά ε, θα πρέπει να είναι το κόστος το ίδιο με το αν έστελνε ευρώ από τη Βαρσοβία στις Βρυξέλλες ή σλότη από τη Βαρσοβία στη Βαρσοβία. Οι μόνε πληρωμέ που δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ διασυνοριακέ είναι αν θέλει να στείλει ένα έμβασμα σε σλότη από τη Σόφια στις Βρυξέλλες. Ε, που είναι πολύ σπάνια περίπτωση και, αφορά ένα πάρα πολύ μικρό κλάσμα όλων των διασυνοριακών πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και ακριβό για τις ίδιες τις τράπεζες να διεκπαιρεώσουν αυτή τη συναλλαγή ε, σήμερα. Άρα θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει πόσο θα κόστιζε κάτι τέτοιο και μετά με χαρά να καλύψουμε ε, ότι θέλετε και αυτό το μικρό κλάσμα όλων των διασυνοριακών πληρωμών. Για τη μετατροπή του νομίσματος και τη διαφάνεια είναι αρκετά τεχνικό αυτό το θέμα και με τις ισοτιμίες και έχει κυκλοφορήσει ένα κείμενο για να απαντήσετε γραπτός έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι εκφράζουμε τις ιδέες μας σωστά για να υπάρξει μεγάλη σαφήνεια για το θέμα, για να προχωρήσουμε έτσι αρκετά γρήγορα. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Και τέλος, για το RTS που ανέφεραν οι πράσινοι και ο κύριος Γκίγολτ, Τώρα το να δώσουμε εντολή στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ε, να εκπονήσει τέτοιο σύστημα για να πλαισιώσει τη μετατροπή. Νομίζω ότι αυτό το παρατραβάει, παρά είναι... Ε, δεν χρειάζεται ένα τέτοιο ρυθμιστικό μέτρο. Και η μόνη ομάδα που θέλησε να παραμείνει αυτό στο κείμενο ήταν η πράσινη. Και στις συζητήσεις μας ακόμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τελευταίες εβδομάδες έχουν εγκαταλείψει και οι ίδιοι αυτή την ιδέα. Και η πλειονότητα των ενδιαφερομένων που συνάντησα, για να μην πω όλοι, ε, συμφωνούσαν σε αυτό. Αν υπήρχε ένα σημείο στο οποίο να συμφωνούσαν ήταν αυτό. Πάντως υπάρχει ευρία υποστήριξη να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο. Σας ευχαριστώ προς το παρόν και Προσβλέπω στην ε, μελλοντική συνεργασία με τους Κιώδης. Ευχαριστώ πολύ. Το χρονοδιάγραμμα μόνο. Συζήτηση των τροπολογιών στις 9 το μηνό, σήμερα δηλαδή. Θα ψηφίσουμε στις 5 Νοεμβρίου ε, στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια, μάλλον τον Νοέμβριο. Κλείνει λοιπόν η πρωινή συνεδρία σε ραντεβού στις 2.30 συζήτηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Προσέξτε, ψάξτε το όνομά σας γιατί αλλάζει η διάταξη των εδράνων. Καλή σας όρεξη και θα τα πούμε μετά. Ευχαριστώ.